Please, if you may, if we all may have your silence. Αν θέλετε να ησυχάσουμε για να ξεκινήσουμε παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας καλωσορίζω εκ νέου. Καλό βράδυ σε όλους. Να ξεκινήσουμε έχουμε δυόμιση ώρες αν τα καταφέρουμε και νωρίτερα, καλύτερα θα είναι για άλλους. Λοιπόν, να εγκρίνουμε το σχέδιο της ημεζίας διατάξεως. Υπάρχει μία αλλαγή πέραν της... Ε, μάλλον είχαμε μία ψήφο μετά τη συνάντηση των συντονιστών υπό το 6-2 σχέδιο προγράμματος και κατάλογος εμπειρογνωμόνων για την ελευθερία του τύπου, της ελευθερίας έκφρασης και τα μηνύματα μίσους online κτλ. Και το σημείο 3 αν, ανεβλήθη η εκλογή τρίτου αντιπροέδρου. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, δεν ξέρω αν έχουμε αντιρρήσεις, αν δεν έχουμε, θεωρώ ότι έχουμε γκρίνει, παρακαλώ. Ε, ε πρόεδρε, κάθε φορά να βάλουμε την εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου, ε, εμάς δεν μα βρίσκει σύμφωνο σε αυτό, Πρόεδρε. Θα θέλαμε την επόμενη φορά στου συντονιστές να είναι το σημείο αυτό για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Το σημειώνουμε, λέει ο Προεδρο. Λοιπόν, τώρα ανακοινώσει. Έτσι. This is an There languages, but Estonian, Latvian, Maltese. Έχουμε όλες τις γλώσσες εκτός εστονικών, λετονικών, Ιρλανδικών και Ουγγρικών τα οποία μπορείτε να μιλάτε αλλά όχι και να ακούτε. Έχουμε λοιπόν τις συστάσεις των συντονιστών να εγκρίνουμε πρώτα απ' όλα. Οι εισηγητές Πίτερ Βίνανοφ για τη Λευκορωσία για τους ε, διαμένοντες χωρίς άδεια παραμονής. Το εγκρίνουμε. Έχουμε εκτελεστικές και κατεξιοδότητες συμπράξεις Τουλάχιστον δύο, λέει ο πρόεδρος. Κατ' εξοδότηση. Ο κανονισμό που τροποποιεί τον κανονισμό για το εσωτερικό Ταμείο ασφαλεία. Αυτό έχει διαβιβαστεί σε όλα τα μέλη της ΛΥΜΠΕ μέσω email. Υπάρχει εσωτερική προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων. 29 Οκτωβρίου το μεσημέρι άλλη μία κατεξιοδότηση ο κανονισμός που συστήνει το Ταμείο για το Άσυλο για τη Μετανάστευση έχει δυναμηθεί επίσης με εσωτερική προθεσμία 29 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Έχουμε και δύο εκτελεστικές το παράρτημα της απόφασης της Επιτροπής για τους τεχνικούς κανόνες, για τη σύνδεση δεδομένων από διάφορα στήματα πληροφορικής και αυτό έχει διαβιβαστεί στα μέλη της ΛΥΜΠΕ μέσω newsletter στις 15 Οκτωβρίου στις 18 Οκτωβρίου μάλλον έχουμε και εδώ 29 Οκτωβρίου προθεσμία Επίσης έχουμε το European Search Portal, τη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης, με προθεσμία για αντιρρήσεις 30 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Και τώρα έχουμε κάποιες πληροφορίες που είναι το πρώτο ουσιαστικό σημείο για σήμερα. Η πρώτη για τη συνάντηση των συντονιστών 6-2 στην οποία αναφέρθηκα και για την αλλαγή του σχεδίου προγράμματος και του καταλόγου εμπειρογνωμόνου για την ακρόαση ΛΥΜΠΕ για την ελευθερία τύπου, ελευθερία έκφρασης, μηνύματα μίσους online και offline, λέει ο πρόεδρος. Ε, η πλειοψηφία των συντονιστών έχουν εγκρίνει το σχέδιο του προγράμματος για το πλαίσιο αυτό, το οποίο προλαμβάνει ο πρόεδρος. Και τώρα από εμάς εξαρτάται να ψηφίσουμε, να εγκρίνουμε δηλαδή τη σύσταση των συντονιστών. Η διαδικασία της ψήφου θα έχει ως εξή. Αν συμφωνείτε με τις συστάσεις των συντονιστών για το σχέδιο του προγράμματος και τον κατάλογο των υπηρεγόμενων και το εγκρίνετε, θα ψηφίσετε συν. Αν είστε κατά για το σχέδιο προγράμματος και τον κατάλογο των υπηρεγόμενων, θα, θα ψηφίσετε μείον. Κατανοητό. Ένα λεπτό, κυρία Ταρδίνο. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήθελα να εξηγήσω σαφέστερα, λέει η κυρία Ταρντίνο, τον λόγο για τον οποίο το ζητήσαμε αυτό. Κάποιες από τις προτάσεις μας δεν συμπεριλήφθησαν στο ελληνικό σχέδιο προγραμμάτων όπως το ενέκριναν οι συντονιστές. Δεν είναι πρώτη φορά. Λυπούμεθα για την έλλειψη δημοκρατικών κανόνων ε, για τους οποίους πάντοτε μιλούμε και ήθελα να θυμίσω ότι η ομάδα μας με τους 73 βουλευτές έχει, είναι το 10% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκπροσωπεί και επομένως είναι η βούληση πολλών ευρωβουλευτών και έκφραση πολλών πάρα πολλών ψήφων των πολιτών. Εδώ χρειάζεται μια ισότητα μεταχείρισης υπό την ε, σωστή αριθμητική αναλογία. Χρειαζόμαστε έναν ομιλητή για κάθε δέκα που επιλέγονται. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα και υποχρέωση θα έλεγα. Ε, η δημοκρατία είναι κάτι στο οποίο αναφερόμαστε συχνά, αλλά με το λάθος τρόπο. Ο Πρόεδρος, ε, ευχαριστώ. Ακούσατε τους ID Όσοι είστε λοιπόν υπέρ τη είστε των συντονιστών να ψηφίσετε συν, όσοι είστε κατά και είστε επομένω υπέρ τη πρώτη του ID, θα ψηφίσετε μείον. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. No, it doesn't work. doesn't work. Eh? No. Now the vote is closed. Πέρασε. Λοιπόν, εγκρίναμε τη σύσταση. Πρέπει να κάνουμε δεύτερη ψηφοφορία, αλλά έχω πρόβλημα, λέει ο πρόεδρο. Διότι έχουμε μία πρόταση ψηφίσματο τη οποία την χάνει να είμαι εισηγητή, αλλά η κάρτα μου δεν δουλεύει. Άρα θα υπολογίσω τον εαυτό μου και με συγχωρείτε εκ των προτέρων Ναι, γι' αυτό δεν δουλεύει, λέει ο πρόεδρος, σε κάτι που ελέγχθη εκτός μικροφώνου και δεν το ακούσαμε. Θα σηκώσω λοιπόν το χέρι μου, ώστε να με μετρήσετε και εμένα. No, no, no, I mean, yes, esta, no funciona. Es el último mandato. Well, the point is search and rescue είναι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης ή στη Μεσόγειο. Κατόπιν ε, προφορικών ερωτημάτων, προφορικού ερωτήματος μάλλον, που είχαμε εδώ, Στρασβούργο, ψήφισμα για θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για όλους μας με τους θανάτους στη Μεσόγειο και όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα. Παρακαλώ να ψηφίσουμε διαδικαστικό. Ποιος? Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, εδώ είμαι. Ε. Μας το στείλατε το ψήφισμα στα αγγλικά για μία ακόμα φορά. Δεν είχαμε μετάφραση. Λυπούμε. Την τελευταία φορά είχατε πει ότι αυτό είναι όλος εξαιρετικό. Σας είχε γίνει η παρατήρηση, το σχόλιο. Σας ζητώ πραγματικά να σεβόμαστε τις γλώσσες των χωρών. Κάνετε μία προσπάθεια, αν δεν θέλετε να αποχωρούμε από την αίθουσα επικειμένων που δεν είναι μεταφρασμένα στη γλώσσα μας στη μητρική μας γλώσσα, λέει ο Ναι, αυτό το αποφάσισαν στους συντονιστέ, λέει ο πρόεδρος, ε, και ε, αυτοί αποφάσισαν, αυτοί αποφασίζουν. Ζητώ συγγνώμη και από ό,τι κατάλαβα οι μεταφράσεις θα είναι έτοιμες εντός της εβδομάδος, εντός της τρεχούσης εβδομάδας. Σε μια-δυο μέρες θα είναι έτοιμες, σε όλες τις γλώσσες. Αλλά σήμερα για την ψήφο. Έτσι αποφάσισαν οι συντονιστές. Ε, ναι, αλλά πρόεδρε μου είπαν ότι δεν, τέτοια συμφωνία δεν είχε δοθεί στους συντονιστές. Δεν είχε δοθεί. Έτσι μου είπαν, λέει ο πρόεδρος. Κάποιος άλλος έχει ζητήσει το λόγο. Α, για διαδικαστικό. Είναι πραγματικά διαδικαστικό. για να δούμε. Ένα λεπτό. Ναι, θέλω να αναβάλουμε ε, για την ψηφοφορία αυτή, γιατί οι συντονιστές δεν μπορούν να, να ε, παραβούν τα δικαιώματα των ευρωβουλευτών. Είναι θεμελιώδες το, το ερώτημα του αν θα υπάρχει το ψήφισμα σε όλες τις γλώσσε γλώσσες ή έστω στις μεγαλύτερε γλώσσες. Έτσι, έτσι δουλεύουμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Αν δεν εξασφαλίζεται η μετάφραση, αυτό σημαίνει ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα των ευρωβουλευτών. κοιτάξτε, έτσι έχουν τα πράγματα, κύριε Ραντζέλ. ότι the coordinators Have no Κοιτάξτε, οι συντονιστέ δεν έχουν καμία δικαιοδοσία και εξουσιοδότηση να τροποποιούν τι βασικέ αρχέ και τα βασικά δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν να αλλοιώνουν την ίδια τη φύση τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μια πολύγλωση κοινότητα. Επομένω, λέω το εξή. Δέχομαι ότι για λόγους ε, διευκόλυνσης των εργασιών μπορεί να έχουμε μία ή δύο γλώσσες, ε, αλλά στις επίσημες επιτροπές ε, και στην Ολομέλεια θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ο καθένας την εκδοχή, τη γλωσσική του. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να διαβάσω έξι γλώσσες, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα, είναι θέμα αρχή. Because... Παρ' όλα αυτά, λέει ο πρόεδρο, πρέπει οπωσδήποτε να περάσουμε στην ψηφοφορία, καθότι έχει ληφθεί η σχετική απόφαση από του ε, και βάσει των, ε, του κανονισμού λειτουργία του Σώματο έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μια τέτοια απόφαση. Αποφασίστηκε λοιπόν έτσι από του συντονιστέ και επομένω δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία.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 No, it's, it's, it's the coordinators. It's decision. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος, είναι απόφαση των συντονιστών. Let's go. Και άρα προχωράμε. Αιτιολογική σκέψη D, άρχεται η ψηφοφορία. Υπέρ. Υπέρ. Είμαστε στην ιδεολογική σκέψη D. Drink. Ηλεκτρονικά δεν ψηφίζουμε. Α, ναι, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά έχετε δίκιο, άρα όχι υπέρ, κατά κλπ. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν, πάντα επί τη αιτιολικής σκέψη D. ECR plus one. ECR plus one too many. Υπάρχει ένα ECR παραπάνω από ό,τι πρέπει. Okay. So now they should... eh? One should uh, redo. Okay, we can close. Close. It's been withdrawn. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περανάμε στην αιτιολογική σκέψη J, άρχεται η ψηφοφορία. Αιτιολογική σκέψη J, άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρα τη ψηφοφορία. Ε, ε, το ΕΛΚ έχει μια παραπάνω ψήφο. Να αποσυρθεί κάποιο, παρακαλώ. Closed. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη L. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Αγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα την παράγραφο 2, λέει ο Πρόεδρος. Έκανα λάθος όμως. Διορθώνει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε την εντολική σκέψη «ΟΟΥ». Άρχεται η ψηφοφορία. Closed. Πέρας της ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Τώρα όμως ψηφίζουμε την παράγραφο 2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Διονομαστικής κλίσεως μετά από αίτημα του ΕΛΚ. Παράγραφος 4, ονομαστική ψηφοφορία λοιπόν. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Ψηφίζουμε. Πάλι διονομαστικής κλίσεως άρχεται. Closed. Ναι. Εγκρίνεται. Ναι, εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Άρχεται. Get me there. On favor. Closed. Πέρας. Και εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Άρχεται. Πάλι διονομαστικής κλήσεως. Πέρας. It's rejected. Απερίφθη. Παράγραφος 10. Διονομαστικής κλήσεως. Now it's closed. Πέρασε. Απερίφθη. Παράγραφος παριθμό 13. Πάντα διονομαστικής κλήσεως άρχεται η ψηφοφορία. Closed. Now it's a... Πέρας και εγκρίνεται. Παράγραφος 14. Άρχεται. Now closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 16. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Παράγραφος 20. Άρχεται. Παράγραφος 19 διορθώνει ο Πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Παράγραφος 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. Και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία διονομαστικής κλίσεως ε, επί του τροποποιηθέντος κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Now, we welcome to this podium. Και τώρα, σας παρακαλώ ησυχία. Συντομεύετε. Antoine, ¿puedes, puedes pedirle a, a Carmen? Please, no interruption. We welcome here. Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, Παρακαλώ ησυχία. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Συντομεύετε και σας παρακαλώ να κάνουμε ησυχία για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Έχουμε μία ώρα μπροστά μα και θα την αφιερώσουμε σε μια ανταλλαγή απόψε με την κυρία Ντούνια Μιγιάτοβιτς, η οποία είναι Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Είναι μεγάλη μα τιμή και μεγάλη μα χαρά που σας καλωσορίζουμε εδώ, κυρία Επίτροπε. Μια εξαιρετικά σημαντική υπηρεσία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ανέλαβε τα καθήκοντά τη τον Απρίλιο του 2018, πάνω από ένα χρόνο. Και εργάζεται ε, πάνω σε μια σειρά ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά και για εμάς, όπως μετανάστευση, άσυλο, ελευθερία του τύπου. Και είμαι πολύ χαρούμενος που επιτέλους τα καταφέραμε να την υποδεχτούμε εδώ για μια ανταλλαγή απόψεων. Εδώ, στο Στρασβούργο στην κοινή μας έδρα, την κοινή έδρα των δύο θεσμικών μας οργάνων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα την ακούσουμε, στη συνέχεια θα ακούσουμε τους συντονιστέ και στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μας για ερωτήσεις, παρατηρήσεις που θα θελήσουν να απευθύνουν στην Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κυρία Μιγιάτοβιτς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Please. Silence. Παρακαλώ ησυχία. Ας σεβαστούμε την προσκεκλημένη μας, που έχει ήδη λάβει το λόγο. Σας παρακαλώ ησυχία για να ακούσουμε με προσοχή τα όσα έχει να μας πει η Επίτροπος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, είναι χαρά μου και τιμή μου που έχουμε αυτή την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων πάνω στα ζητήματα που εσείς ζητήσατε και που σας ενδιαφέρουν όλος ιδιαίτερος. Έχω πολύ τακτικές επαφές με πολλούς από εσάς και στην προηγούμενη ε, ιδιότητά μου είχα τη δυνατότητα να ανταλλάξω απόψεις με πολλούς από εσάς για ζητήματα που άπτονται των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή την πολύ σημαντική έναρξη της συνεργασίας με το επιτελείο μου πάνω σε μια σειρά πολύ σημαντικά ζητήματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μετανάστευση και την ελευθερία έκφρασης. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη, από σεβασμό προς τον χρόνο σας, αλλά και για να σας δώσω τη δυνατότητα να μου απευθύνετε ερωτήματα, γιατί είναι εξαιρετική η ευκαιρία αυτή και για εσάς να μου απευθύνετε τυχόν ερωτήματα που έχετε. Ζούμε σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ έχω αναλάβει τα καθήκοντά μου εδώ και 18 μήνες και έχω παρατηρήσει πολύ ανησυχητικές τάσεις σε αρκετά μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων ε, που, ορισμένων μάλλον, που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που έχουμε αυτή την ευκαιρία και ελπίζω να συνεχιστεί η τακτική αυτή, η πρακτική αυτή η τακτικά. Θα σταθώ εν συντομία στο ζήτημα της μετανάστευσης ε, και πιο συγκεκριμένα σε κάποια ζητήματα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι η μεταχείριση των μεταναστών είναι η λιδία λήθος ε, για, τα, για τον σεβασμό από πλευράς κρατών μελών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσον αφορά την νομοθεσία, η ανυπαρκή ε, νομοθεσία ή η έλλειψη μέτρων ένταξης ε, έχουν δημιουργήσει ένα πολιτικό χάος. Και η ανταπόκριση σε αυτό το χάος πολύ συχνά είναι πιο περιοριστικές πολιτικές και πιο περιοριστικοί νόμοι και κανόνες. Και λόγω παρά την φθήνουσα, τον φθήνοντα αριθμό ε, άφηξης μεταναστών βάσει των στατιστικών στοιχείων που έχουμε στην Ευρώπη, αυτό που εντοπίζουμε, που θεωρώ ότι είναι πολύ ανησυχητικό, είναι μια ρητορική η οποία δεν είναι εκείνη που θα θέλαμε να ακούμε σε δημοκρατικά πολετεύματα. Όταν γίνονται στόχος ε, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και πιο συγκεκριμένα ομάδες που δεν έχουν τη δυνατότητα και να, να απαντήσουν σε αυτού του είδους τη ρητορική πολλές ε, κυβερνήσεις, μεταξύ αυτών ε, ε, και πολλές κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν καταφέρει να παράσχουν βασικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις σε μετανάστες και ετούντες άσυλο. Μάλιστα θεσπίζοντας μειοπική νομοθεσία, όπως είναι η περιοριστική νόμη για την επανένωση των οικογενειών, η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και η, ε, το, ε, το, το, να καθίσταται πιο δύσκολη η πρόσβαση σε, κοινωνική, σε κοινωνικά επιδόματα. Ελπίζω να είδατε το εγχειρίδιο για την Μεσόγειο που διενεμήθηκε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασης που επικρατεί στη Μεσόγειο ε, στον τομέα της μετανάστευσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξίζει της προσοχής μας. Η σύσταση που περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο αυτό αποτελεί ένα πρώτο έγγραφο όπου προσπαθώ να ε, σταθώ και να αναδείξω ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίω ε, τη κατάσταση των μεταναστών στην Ευρώπη. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε πέντε συγκεκριμένου τομεί δράση που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικοί για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε. Πρώτον, θέλω να αναφέρω την αποτελεσματική έρευνα και διάσωση. Αυτή απαιτεί την ε, ενισχυμένη και βελτιωμένη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων αρχών. Δεύτερον, έγκαιρη, έγκαιρη ε, ασφαλής αποβίβαση. Θα πρέπει οι διασωθέντες να αποβιβάζονται με ασφαλή τρόπο. Αυτό βεβαίω ε, θα γινόταν σε έναν ιδανικό κόσμο. Ξέρω ότι ο κόσμο μα δεν είναι ιδανικό. Ταυτόχρονα όμω πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι και αφοσιωμένοι στι ε, θεμελιώδει αξίε μα και τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Επίσης, ε, θα πρέπει να γίνεται σεβαστή η άρνηση καπετάνιων για την παράδοση μεταναστών όταν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του. Λοιπόν, η, η αποβίβαση είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι συζητήσει που ξεκίνησαν στην ε, Μάλτα εμφανίζονταν, ε, εμφανίζονται να πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση. Είναι μια αρχή, αν θέλετε. Παρακολουθούμε στην Α. Χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια ε, ως προς το πώ θα λειτουργήσει ο μηχανισμό που θα, θα θεσπιστεί και τι είδους εχέγγυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα υπάρχουν. Επίση, εξακολουθώ να έχω κάποιε αμφιβολίε σχετικά με, άλλες, ε, με άλλα τμήματα τη συμφωνία που ε, δείχνει να ε, ενισχύει τη συνεργασία με τρίτες χώρες όσον αφορά την πρόληψη των αφήξεων. Και εδώ φτάνουμε στον τρίτο τομέα, όπου χρειάζεται περισσότερη δράση. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα ε, αναγκαία εχέγγυα στη συνεργασία μας με τρίτες χώρες. Καταλαβαίνω ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά χρειάζεται να έχουν μορφές διεθνούς συνεργασίας όσον αφορά την μετανάστευση. Ωστόσο, μια τέτοια συνεργασία πολύ συχνά δεν διαθέτει ε, τα απαραίτητα στοιχεία διαφάνειας και λογοδοσίας. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να συμβάλλουν στην παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαίνουν σε τρίτες χώρες. Οι αποτρόπες, ε, ε, τα αποτρόπαια αποτελέσματα από τις κρατήσεις της Λιβιακής Ακτοφυλακής είναι πλέον αποδεδειγμένο ε, γεγονός. Γι' αυτό και χρειάζεται να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Τέταρτο τομέα είναι η παροχή ασφαλών και νόμιμων οδών. Αυτό απαιτεί την ε, ενισχυμένη συνεργασία σε μηχανισμούς και συστήματα επανεγκατάστασης μεταναστών, ανθρωπιστικές θεωρήσεις, ε, συστήματα και μηχανισμούς χρηματοδότησης και εξασφάλιση γρήγορης και ασφαλούς επανένωσης οικογενειών. Επίσης, είναι απολύτω ζωτική σημασία η σωστή και καλή συνεργασία με ε, μη κυβερνητικέ οργανώσει. Δυστυχώ το αντίθετο έχει γίνει. Η συκοφάντηση ε, αυτών των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι ο κανόνα. Αυτό το παρατηρώ από την αρχή τη ε, θητείας μου και δυστυχώ δεν φαίνεται να σταματά αυτή η τάση. Εγώ εκτιμώ τι εργασίε σα για την αποποινικοποίηση των δραστηριοτήτων των μη κυβερνητικών οργανώσεων που βοηθούν μετανάστες είναι σημαντικό στο μέσο συνεργασία. Τώρα, να σταθώ λίγο και στι ε, συνθήκε υποδοχή που εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ ανησυχητικέ σε πολλά κράτη-μέλη. Ιδίω στην Ελλάδα η κατάσταση είναι εξαιρετικά πιεστική. Δεδομένη τη ε, τρέχουσα κατάσταση, ε, ε, την επόμενη εβδομάδα θα ξαναεπισκεφτώ την ε, Ελλάδα. Είχα πάει και πέρσι τον Ιούνιο, θα πάω και στη Σάμο αλλά και στην πυροτική χώρα. Και θα δημοσιεύσω τα ευρήματά μου και βεβαίω με χαρά ε, θα επανέλθω εδώ στην Επιτροπή σα για να ξανασυζητήσουμε το ζήτημα. Βεβαίω η Ελλάδα δεν είναι η μόνη τη όσον αφορά τι συνθήκε διαβίωση που κρατούνται σε ανεπαρκεί εγκαταστάσει. Και αντί να σα δώσω έναν κατάλογο χωρών, θέλω να σταθώ σε ορισμένε γενικέ παρατηρήσει. Σε κάποιε περιπτώσει ο αριθμό των αφήξεων πράγματι ήταν πολύ υψηλό, προ, προκαλώντα προβλήματα στα κράτη-μέλη που του υποδέχονταν. Όμω η ευρωπαϊκή ανταπόκριση ε, μια διαχειρίσιμη κατάσταση την ε, έκανε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Αυτό οφείλεται σε έλλειψη επενδύσεων σε συστήματα υποδοχής και στην αποτυχία των κρατών μελών να προχωρήσουν σε έναν δίκαιο επιμερισμό των βαρών. Η συνολική στάση σε ορισμένα κράτη-μέλη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται από απροθυμία να δοθεί η ε, αναγκαία απάντηση. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε δεν είναι ένα ε, πρόβλημα μόνο ενός κράτους μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και όταν λέω ευρωπαϊκό, δεν ε, αναφέρομαι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ την Ευρώπη ως Ήπειρο. Οι επενδύσεις λοιπόν στην υποδοχή και στην εκπαίδευση εκείνων που δικαιούνται να μείνουν εδώ Επίση δεν ανταποκρίνονται στι ανάγκε. Και αυτό θα ήταν ο μόνο τρόπο για να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να διαχειριστεί τι μελλοντικέ μεταναστευτικέ ροέ με τρόπο που θα διασφαλίζει ε, τα δικαιώματα και των ίδιων των μεταναστών και των κοινοτήτων υποδοχή του. Υπάρχουν και παράνομε απελάσεις ω μέτρο για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών καθώ και το θέμα τη προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων. σω θα μπορούσαμε να σταθούμε σε αυτό το ζήτημα και στη συζήτηση που θα έχουμε αλλά και κάποια άλλη στιγμή ενδεχομένως. Το δεύτερο θέμα, στο οποίο θέλω να σταθώ εν συντομία, ε, σχετίζεται με την ελευθερία του τύπου. Από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχω αφιερώσει μεγάλο χρόνο, πολύ χρόνο μάλλον, στην ε, προστασία της ελευθερίας έκφρασης και του τύπου, ιδίως στην προστασία της ασφάλειας των ε, δημοσιογράφων. Πριν από λίγες μέρες εξέδωσα μια ε, ανακοίνωση για τα δύο χρόνια από την αποτρόπαια δολοφονία της ε, Δάφνης Γαλίτσια στην Μάλτα. Ακόμη δυστυχώς δεν έχουμε ε, καταλήξει σε συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα όσον αφορά τη διαλεύκανση αυτού του αποτρόπιου εγκλήματος. Τα κράτη-μέλη έχουν ε, ισχυρά εχέγγυα ε, για την προστασία των δημοσιογράφων. Η ελευθερία του τύπου κατοχυρώνεται και στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και στις εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Οπότε όταν μιλάμε για ψηφίσματα, για νόμους, ε, είμαστε καταπληκτικοί, μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Όταν όμως μιλάμε για την εφαρμογή, ε, και το τι συμβαίνει στην πράξη, τότε πραγματικά ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη συμμόρφωση με του κανόνε αυτού. Πολλά πρέπει να γίνουν αυτά για να μετωσιωθούν αυτά τα πρότυπα και στην ε, πράξη. Όσον αφορά τη Σλοβακική Δημοκρατία, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν κάποια απτά αποτελέσματα όσον αφορά την έρευνα ενό άλλου αποτρόπου εγκλήματο που συνέβη στην Σλοβακία, την δολοφονία του νερού δημοσιογράφου και τη συντρόφου του πλέον η ε, ηθική και φυσική αυτούργοι έχουν συρθεί ε, ενώπιον της δικαιοσύνης και θα αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του νόμου. Ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του τύπου και την προστασία και την ασφάλεια των δημοσιογράφων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει πραγματικά να δούμε κατάματα την πραγματικότητα. Εδώ και δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, ένας χώρος, μια περιφέρεια του κόσμου ασφαλής, που παρήχε ένα περιβάλλον όπου ένας δημοσιογράφος πραγματικά μπορούσε να ε, εκτελεί την εργασία του ε, με ελευθερία και ασφάλεια. Δολοφονίες λοιπόν που έγιναν τα τελευταία χρόνια στη Σλοβακία, Μάλτα αλλά και στην ε, Βουλγαρία δυστυχώς βλέπουμε να χαράσουν έναν δρόμο για τον οποίο καθόλου περήφανοι δεν πρέπει να είμαστε. Γι' αυτό και δεν πρέπει να επιτρέψουμε την ασυλία και την ατιμορρησία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό εξ αυτού του λόγου εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ εντό εντός τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να διερευνηθούν ε, πλήρως τα εγκλήματα αυτά, όχι μερικώς, ε, για να μην δημιουργηθεί ένα άσχημο περιβάλλον ε, στο, για την εργασία των δημοσιογράφων. Συμφωνούμε όλοι ότι το τοξικό αυτό περιβάλλον δηλητηριάζει τη δημοκρατία. Αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί. Επίσης, εργάζομαι σε χώρες που βρίσκονται σε μετάβαση. Εκεί όπου υπάρχουν άνθρωποι που είναι δημοσιογράφοι και εκτελούν την εργασία τους από, από τη φυλακή με συνεχή καταστολή και εκφοβισμό όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τις οικογένειές τους και τους φίλους τους. Αυτά τα προβλήματα ε, δυστυχώς είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν τώρα που οι εθνικισμοί ενισχύονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Διότι όχι μόνο θεωρούν οι εθνικισμοί αυτοί αντίπαλο τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά αξιοποιούν και την θέση εξουσίας που έχουν για να ε, ε, εκφοβήσουν ε, μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους. Αυτό το εχθρικό περιβάλλον δυστυχώς νομιμοποιεί τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων. Στο ρόλο μου ως Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης θέλω να συνεχίσω να δίνω ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Νομίζω ότι τα κράτη πρέπει να ενθαρρυνθούν, να ανταλλάσσουν θετικέ εμπειρίε που υπάρχουν από άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Υπάρχουν κάποια καλά παραδείγματα και θέλω πάντοτε να στέκομαι και σε αυτά. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, όπου πολλοί δημοσιογράφοι είχαν δολοφονηθεί στο παρελθόν και άλλοι πολλοί είχαν αντιμετωπίσει διάφορε απειλέ συμπεριλαμβανομένης και πολύ εχθρικής ε, πολιτικής ρητορική. η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές ε, έχουν καταφέρει εδώ και πολλά χρόνια να προστατεύουν τη ζωή των δημοσιογράφων. Στις κάτω χώρες η εισαγγελία, ε, η αστυνομία, οι δικαστικές αρχές και οι δημοσιογράφοι έχουν καταφέρει να συνάψουν μια συμφωνία για την προστασία των δημοσιογράφων. Αντίστοιχα φαινόμενα υπάρχουν στην Σουηδία. Οπότε υπάρχουν και καλά παραδείγματα. Οι κυβερνήσει επίση θα πρέπει να υποστηρίζουν πρωταβουλίε των, οργανω... των οργανώσεων των δημοσιογράφων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και πανεπιστημιακών φορέων. Ιδίω όσον αφορά την χαρτογράφηση και την ε, αναφορά απειλών κατά δημοσιογράφων, όπου ε, πραγματικά είναι ένας ε, εξαιρετικά, ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για να μπορεί κανείς να προλαμβάνει τέτοιου είδους φαινόμενα και επιθέσεις σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ε, επίσης υπάρχουν δυστυχώς χώρες ε, όπου υπάρχει ε, αστυνομική βία κατά διαδηλωτών. Ιδίω ενάντια στου δημοσιογράφου που καλύπτουν τι διαδηλώσει αυτή, που είναι πολύ συχνά ο πρώτο στόχο. Αυτό πρέπει να αναγνωριστεί και εδώ ε, μιλάμε ακόμη και για κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να κάνουν περισσότερα. Πρέπει να, γίνει περισσότερη, να δοθούν περισσότεροι κύκλοι εκπαίδευση, κατάρτιση σε αστυνομικού αλλά και σε, σε άλλου θεσμικού φορεί και να εξηγείται διαρκώ ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να είναι στόχο τέτοιων φαινομένων. Πολύ ε, πρόσφατα έχω εκδώσει και σχετικές ανακοινώσεις, αλλά θα επανέλθω σε αυτό το ζήτημα. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λοιπόν είναι μια καθημερινή εργασία, ένα καθημερινό καθήκον που ταυτόχρονα συνοδεύεται από ένα μακροπρόθεσμο όραμα. Και εσείς είστε πραγματικά εταίρος μου στην ε, προσπάθεια αυτή. Θέλω να ακούσω τις ερωτήσεις σας και προσβλέπω πραγματικά στην ενισχυμένη και βελτιωμένη συνεργασία μας σε, στα ζητήματα στα οποία στάθηκα εγώ σήμερα, αλλά και για πολλά άλλα ζητήματα, γιατί εγώ ξέρετε στάθηκα μόνο σε κάποια λίγα ζητήματα. Μιλάμε τώρα για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ, των ΛΟΑΤ, τα δικαιώματα του παιδιού, τα δικαιώματα των γυναικών, ε, και πολλά άλλα ζητήματα που βρίσκονται πολύ ψηλά στην ατζέντα μου και που θα παραμείνουν ε, σε αυτήν ως προτεραιότητες. Ε, ευχαριστούμε την κυρία Μιγιάτοβιτς. θα έχουμε ένα γύρο για τους συντονιστές και μετά θα δώσουμε το λόγο στα μέλη για να απευθύνετε τα ερωτήματά σας στην Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, κυρία Μετσόλα, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Μιγιάτοβιτς. Ε, σωστά λέει ότι αυτοί που χρήζουν προστασίες είναι εκείνοι των οποίων πλήττονται περισσότερο ανθρώπινα δικαιώματα και ε, τα χρήματα δεν είναι το παν, αλλά βοηθούν. Έχουμε δει την πίεση να αυξάνεται την ένταση να οξύνεται και είμαστε σε θέση να ίσως να εντοπίσουμε κάποιες βέλτιστες πρακτικές και ίσως να μας πείτε κι εσείς εάν έχετε δυνατότητα λίγα περισσότερα πράγματα για το πώς έχει η κατάσταση στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε επίσης για τη φωνή σας ε, στο θέμα της ελευθερίας του τύπου πάντοτε τοποθετήστε με σαφήνεια για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προτύπων που πρέπει να παρακολουθούνται από τα κράτη-μέλη σχετικά με την προστασία των δημοσιογράφων και των εκπροσώπων του τύπου και προερχόμενοι και από τη Μάλτα ε, νομίζω ότι χρειάζεται δικαιοσύνη για την δολοφονημένη Ντάφνη Γκαλίτσια. η κυβέρνηση του κυρίου Μουσκάτ ε, ε, προσπαθεί να παρουσιάσει το θέμα ως ένα θέμα κομματικής φύσεως και ίσως θα ήταν ε, ακόμη πιο ενδιαφέρον να ακούσει την αλήθεια από εσάς. Επίσης μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η εκτίμησή σας σχετικά με την αντίδραση, την τοποθέτηση της μαλτέζικης κυβέρνησης σχετικά με τη δολοφονία αυτή και τι μπορούμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνουμε ώστε να έχουμε λογοδοσία από τα κρατημέλη. Η κυρία Σίπελ, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη γιατί είμαι σίγουρη ότι και άλλα μέλη θέλουν να υποβάλουν ερωτήσει. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα τη μετανάστευση και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μα αρέσει να λέμε ότι είμαστε ήπειρο όπου τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα υφίστανται και, και ότι είμαστε οι καλύτεροι σε αυτό το επίπεδο. Και επικρίνουμε πολύ συχνά επίσης τις τρίτες χώρες σε αυτά τα θέματα, αλλά κοιτώντα την εσωτερική μας εδώ κατάσταση, ιδιαίτερα σε σχέση με κάποια κέντρα προσφύγων συγκεκριμένα, νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι τραγικό όχι μόνο για τους λαούς μας, αλλά και για την ασφάλειά μας και για τον τρόπο ζωής μας. Εσείς αυτές τις εξελίξεις στο ιστορικό της Ένωσης με κέντρα απολύτως ανίκανα να παραλάβουν και να προστατεύσουν τον υπέρογκο αριθμό των ανθρώπων που δέχονται. Επίσης η προστασία των δημοσιογράφων είναι δύσκολο και απαραίτητο έργο. Ε, ε, εγώ μπορώ περνώντας από το δρόμο να πάρω μια φωτογραφία από ένα βίαιο περιστατικό όπου κάποιος χτυπάει κάποιον άλλον αλλά μπορώ εγώ να γνωρίζω ποιος, είναι, ποιος ήταν ένοχος για το επεισόδιο αυτό, ποιος ευθυνόταν αυτός που είναι στο έδαφος ή ο άλλος. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς περιγράφουμε ένα περιστατικό. Η ελευθερία του τύπου και η ελευθερία της έκφρασης έχουν, έχει και αυτή τα όρια της όταν μειώνουμε την ελευθερία των άλλων ή όταν ρέπουμε προς μηνύματα μίσους και παραπληροφόρηση. Υπό την επιτική γωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης, εσείς πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην Ευρώπη όχι μόνο λόγω των δολοφονιών, αλλά και λόγω γενικώς της δυνατότητας που έχουν δημοσιογράφοι να λειτουργούν σωστά στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και για, τον, ε, για τα όσα μας είπατε, τόσο ξεκάθαρα σήμερα. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ εύκολα με όλα αυτά που είπατε και τις παρατηρήσεις που κάνατε. Το ερώτημα βεβαίως είναι τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Και εδώ τα ερωτήματα είναι δύσκολα και έχω την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολύ αργό ρυθμό, υπερβολικά αργό ρυθμό, αναπτύσσει εργαλεία ε, σύμφωνα με τις ε, αξίες τις οποίες διατυμπανίζουμε ε, και λέμε ότι για τις οποίες νοιαζόμαστε. Ε, όμως, επαναλαμβάνω, όταν μιλάμε για το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ στο Στρασβούργο, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι πολλές ε, χώρες είτε αρνούνται είτε δεν δέχονται να εφαρμόσουν τις αποφάσεις. Τι μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε να αυξηθεί ο σεβασμός απέναντι στις αποφάσεις του δικαστηρίου. Δεύτερον, η Ρωσία ξανά είναι μέλος χωρίς ε, υποσημειώσεις και προϋποθέσεις. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Είναι ξανά μέλος. Τίποτα δεν άλλαξε νομίζω. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, εν πάση περιπτώσει να επαναδιατυπώσω τότε. Ε, ξανά έγινε μέλος ε, η Ρωσία στο Συμβούλιο της Ευρώπης χωρίς ιδιαίτερες προϋποθέσεις. Και κάτι άλλο. Πώς μπορείτε να ορίσετε ή να χαρακτηρίσετε αυτό που κάνει η Τουρκία αυτή τη στιγμή και πιστεύετε ότι υπάρχει και ε, φόβος, κίνδυνος για εθνοκαθάρσεις όπως ορισμένοι ανέφεραν. Έχουμε την ε, αίσθηση επίσης ε, ότι ε, πολλοί κάνουν λόγο για πάρα πολλά ζητήματα, για... Not just did he want to attack the synagogue, ε, τι γίνεται στην ε, Συρία, δηλαδή λένε για τις ε, επιχειρήσεις στο Χαλέπι και τι γίνεται και με τις γυναίκες, με τα δικαιώματα των γυναικών, το φεμινισμό, τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων. Δηλαδή πολύ συζητάμε και πολλής λόγος γίνεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά, αλλά ειδικά για αυτά τα δικαιώματα του σεξουαλικού προσανατολισμού δεν γίνεται πολλής λόγος επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μας είπατε και για την πολύ καλή δουλειά που κάνετε. Ξέρω ότι δουλεύετε και με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και ξέρω πόσο σημαντικό είναι το έργο σας για όλους τους πολίτες των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, συμπεριλαμβανομένων ε, και των ε, παρεμβάσεων που κάνετε που είναι ιδιαίτερα δυναμικές. Ευθύνη και λογοδοσία σε πάρα πολλές περιοχές και σε πάρα πολλά θέματα και μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας και με όλα αυτά που είπατε. Ναι, θα πρέπει να αναλάβουμε ευθύνη και για τις ε, πρόσφυγες και για τους ενδυνάμει πρόσφυγες. Ε, ξέρετε τι γίνεται με τις επαναπροωθήσεις στα σύνορα ε, και ξέρουμε και σε πολλές χώρες αλλά και στην Κορατία και στη Βοσνία Ζεγοβίνη γίνονται τέτοιες κινήσεις. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς στο Συμβούλιο της Ευρώπης έτσι ώστε να καταπολεμήσετε την κατάσταση αυτή. Επίσης πώς μπορείτε να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση με το Συμβούλιο της ε, Ευρώπης έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ε, υλοποίηση, επιβολή των ε, αποφάσεων και κάτι άλλο, η λογοδοσία δεν υπάρχει λογοδοσία, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνη όσον αφορά ε, πρόσφυγες ε, από τρίτες χώρες, οι οποίες όμως είναι χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, συζητήσαμε τα θέματα αυτά και με τους υποψηφίους επιτρόπους αρμοδίους για τα θέματα αυτά που θέλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία με αυτές τις τρίτες χώρες και ρωτούν πώ μπορεί να υπάρξει ε, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ίσως έχετε εσείς κάποιες ιδέες για το πώς μπορούμε να παρακολουθούμε όλη αυτή την κατάσταση περισσότερο, πώς είναι δυνατόν ας πούμε ε, να κάνουμε κάποιες αξιολογήσεις κινδύνου πριν ξεκινήσουν ε, κάποιες διαδικασίες. Θα ήθελα να μου πείτε τις απόψεις σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρτίνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο με την έρευνα και διάσωση και αυτές τις δραστηριότητες γιατί ε, συζητήθηκε και θα ξαναζητήθηκε στην Ολομέλη το θέμα αυτό. Ε, στο Συμβούλιο Υπουργών ΔΕΗ ε, υπήρχαν τρία σημεία της ε, ημερησίας διατάξεως και εκεί εσείς ε, και μεταξύ αυτών και την σύμβαση της Μάλτας και είπατε ότι θα πρέπει όσο γίνεται περισσότερες χώρες να προσυπογράψουν τη συμφωνία αυτή. Τέσσερις ήταν οι αρχικές χώρες και άλλες τρεις οι οποίες φαίνεται να δείχνουν διαθεσιμότητα. Δεν υπήρξε άλλη προσυπογραφή αυτής της συμφωνίας, μια συμφωνία όμως που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως ε, μπλόφα παρά καλό σημείο εκκίνησης ε, και από ό,τι φαίνεται τίποτα δεν θα αλλάξει, ιδίως εάν σκεφτεί κανείς ε, και την τελευταία αποβίβαση με πλοίο μη κυβερνητική οργάνωση στον Τάραντα της Ιταλίας. Επομένω, σα ρωτώ, ποια είναι η άποψή σας για αυτή τη συμφωνία και υπό το φως της συμφωνίας ε, του Συμβουλίου επ' αυτού, ε, ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και επίσης να σας πω ότι κανείς δεν θέλει να θέσει σε αμφισβήτηση τα ανθρώπινα δικαιώματα των αντίων. Εμείς πιστεύουμε ότι αντιθέτως εάν συνεχίσουμε να φέρνουμε μετανάστες στην ε, Ευρώπη, ε, τότε θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Προκατσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις από μένα. Άνθρωποι με μεγαλύτερο κύριος από εμένα, δύο πάπες μάλιστα, είχαν πει ότι προτού να προστατεύσουμε το δικαίωμα προς τη μετανάστευση, οι πλουσιότερες χώρες θα έπρεπε να ασχοληθούν με το δικαίωμα της μη μετανάστευσης. Το δικαίωμα του να μην υποχρεώνεται κανείς να εγκαταλείψει τη χώρα του, να αφήσει τη ζωή του, να διακινδυνεύσει τη ζωή του για να διαβεί τη Μεσόγειο, για παράδειγμα. Εσείς δεν πιστεύετε ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα ώστε να βοηθά τους πληθυσμούς και τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες. Δεύτερον, εγώ είμαι απολύτως πεπισμένος ότι η νόμιμη μετανάστευση είναι απαραίτητη και επομένως πρέπει να ρυθμίζεται. Όμως, δεδομένου του ότι οι οικονομικοί μετανάστες δεν θα μπορέσει μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους εξασφαλίσει στους οικονομικούς μετανάστες αξιοπρε... αξιοπρεπή διαβίωση σε όλους αυτούς που προσέρχονται. Ο επαναπατρισμός λοιπόν είναι παραβίαση των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων. Το να παρεμποδίσουμε να εισέλθουν οι μετανάστες στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται ότι είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυρία Ernst. Ευχαριστώ. Καταρχά για το γεγονός ότι βρίσκεστε εδώ και πραγματικά σε πολλά ζητήματα ε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εδώ, εδώ πίσω. Στην τελευταία σειρά με βάλανε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πραγματικά μιλήσατε μέσα από την ε, καρδιά μου ε, και νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να δούμε το θέμα του πώς θα προχωρήσουμε στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν δύο είδη μεταχείριση: Τα ανθρώπινα δικαιώματα που ισχύουν λίγο πολύ εδώ στην Ευρώπη, αλλά όχι για εκείνου που έρχονται στην Ευρώπη. Και εκεί πολλέ φορέ μα είναι αδιάφορο το τι συμβαίνει. Μπορεί να λέμε διάφορα ωραία λόγια, αλλά σε τελική ανάλυση αυτά που συμβαίνουν με του μετανάστες στα εξωτερικά μα ε, σύγχρονα, είτε στη Μεσόγειο, είτε στην ε, Λιβύη, είτε ακόμη και στην υπηρετική Ευρώπη, ε, πραγματικά περνάει τελείω αδιάφορο σε πάρα πολλού που μπορεί ακόμη και να μιλάνε για το ζήτημα. Νομίζω ότι κάποιες φορές έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε ένα σε ένα τροχό ε, του χάμστερ. Ότι λέμε και ξαναλέμε τα ίδια πράγματα, προτείνουμε και ξαναπροτείνουμε τα ίδια πράγματα χωρίς ποτέ να αλλάζει, να κάτι. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ε, απογοητευμένη που σήμερα στην Ολομέλεια απερίφθη το ζήτημα, το, το ζήτημα της κατάστασης που επικρατεί στο Ούτσιακ στην ε, Βόρεια ε, Βοσνία για το ότι δεν καταφέραμε να έρθουμε σε συμφωνία για να υποβληθεί το ε, ψήφισμα δεν μπορώ να το εξηγήσω ούτε στον εαυτό μου ούτε σε κάποιον άλλον. Ε, πραγματικά το ζήτημα είναι ε, ζήτημα ζωής και θανάτου. Δεν υπάρχει τροφή και νερό. Ξέρετε πόσο έκτακτη είναι η κατάσταση εκεί και δεν ε, θα μιλήσουμε ούτε δυστυχώς εδώ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενώ τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε. Αυτά με ανησυχούν εμένα. Εσείς ποια είναι η γνώμη σας, πώς, μπορεί, ε, ε, πώς μπορούν οι πολιτικοί ταγοί να ε, προχωρήσουν. Και το άλλο ζήτημα βεβαίως που με απασχολεί είναι η συμφωνία με την Τουρκία. Η αντιμετώπιση της Τουρκίας και στο πλαίσιο της τρέχουσας συγκρίας. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται τη συμφωνία αυτή διαρκώς για να ασκεί πίεση προς την Ευρώπη παρά το γεγονός ότι ήδη δεν ε, εφαρμόζεται. 23.000 Σύριοι έχουν ε, απελαθεί από την Τουρκία ε, στη Συρία. Ίσως θα μπορούσατε κι εσείς να μας πείτε τη δική σας γνώμη, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να ενισχύσουμε την ε, πολιτική μας θέση. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ακούσατε τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν δεν έχετε αντίρρηση, θα έλεγα να ε, συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για μισή ώρα, να ακούσουμε μάλλον πρώτα όλα τα μέλη της Επιτροπής και συνέχεια να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε συνολικά σε όλους. Οπότε, αν δεν έχετε αντίρρηση, να δώσω το λόγο τώρα στα μέλη της Επιτροπής μας. Η κυρία Νεβιτσένε από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημά μου αφορά μια πιθανή επίσκεψη της Επιτρόπου στην Κρυμαία που έχει ε, προσαρτηθεί παρανόμως από την ε, Ρωσία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ανύπαρκτα στην Κρυμαία. Η Ρωσία έχει καταργήσει την ελευθερία του τύπου και της έκφρασης. Ε, όσοι επικρίνουν την κατοχή αυτή δολοφονούνται και εγώ προσωπικά έχω βιωματική εμπειρία από αυτό και ξέρω ότι ε, οι αξίες δεν είναι σημαντικές σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που θέλουν οι άνθρωποι είναι κάποιος να τους υπερασπιστεί ε, απέναντι σε αυτές τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις επιθέσεις που δέχονται. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσουμε ότι η πολιτική μη αναγνώρισης και κυρώσεων μπορεί να αλλάξει στην τρέχουσα συγκυρία ότι μπορούμε να μιλούμε με υπηρότερου όρους για την κατοχή, για την παραβίαση ανθρωπινών δικαιωμάτων ή ότι υπάρχει ποτέ περίπτωση να αναγνωρίσουμε το status quo στην ε, Κρυμαία ε, για, με αντάλλαγμα τον διάλογο στον Ντομπά ή την εφαρμογή τη συμφωνίας του Μίνσκ. Η επανεισδοχή τη Ρωσία στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη μπορεί επίση να δημιουργήσει ερωτήματα για το αν οι θεμελιώδει αξίε τελικά ε, είναι αντικείμενο προ υπεράσπιση ή ε, εξακολουθούμε να τι ε, υπερασπιζόμαστε. Κυρία Πίτροπε, εσεί σχεδιάζετε να κάνετε κάποια επίσκεψη στην Κρυμαία. Ε, έχετε έρθει σε επαφή με τις Ουκρανικές αρχές και κατά τη γνώμη σας υπό ποιους όρους θα μπορούσε μια τέτοια επίσκεψη να γίνει στην Κρυμαία χωρίς να θεωρηθεί ότι αυτό ε, αποτελεί αναγνώριση του status quo ή ότι η διεθνής κοινότητα με κάποιον τρόπο ε, αναγνωρίζει την εξουσία και την αρχή της Ρωσίας στην Κρυμαία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, ίσως να γνωρίζετε ότι το Πολωνικό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται σχέδιο νομοσχεδίου για κυρώσεις, ποινές, ποινικέ κυρώσεις μάλιστα, ε, για αδικήματα κατά ανηλίκων, κάτω των 18 ετών, σεξουαλικών αδικημάτων κατάχρησης, το οποίο υποχρεώνει όλα τα μέρη, τους συνυπογράφοντες δηλαδή, να αναλάβουν όλα τα νομοθετικά μέτρα εκείνα που είναι απαραίτητα ώστε τα παιδιά στην ε, πρωτοβάθμια εκπαίδευση να λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με τα κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης ε, που μπορούν να υποστούν. Η Πολωνία είναι χώρα που έχει υπογράψει τη σύμβαση και επομένως η... εσείς θεωρείτε ότι αυτή η ενημέρωση που θα μπορούσε να παρέχεται σε ανήλικα παιδιά δεν θα παραβίαζε τη σύμβαση. Η κυρία Τζουριάνο. Σας ευχαριστώ Επίτροπε, ευχαριστούμε για το μήνυμά σας που αποστέλλετε που αποστήλατε μάλλον ε, για το συνέδριο, στα πλαίσια του συνεδρίου που είχαμε για την ε, προάσπιση της ελευθερίας του τύπου και έκφρασης. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την προστασία αυτή που θα πρέπει να παρέχουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις δημοσιογράφους από απειλές, καταχρήσεις και παρεμβολές, ήθελα να ακούσω την ιδέα σας, τις ιδέες σας σχετικά με το πώς καλύτερα θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Είναι επίγον να λάβουμε μέτρα και χρηματοδοτικά μέτρα προκειμένου να υπερασπιστούμε τους εκπροσώπους της ελευθερίας έκφρασης, δηλαδή τους δημοσιογράφους. Ήθελα να ακούσω τις ιδέες σας επ' αυτού. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο για την τοποθέτησή της ε, σχετικά με κάποιες ε, δηλώσεις του Μαΐου που δυστυχώς είναι πρωτοσέλιδα στον τύπο που αναφέρονταν στην... διακόπτουν την ομιλήτρια αλλά δεν ακούμε. Κάτι λέγεται εκτός μικροφώνου. Μάλλον δεν έγινε κατανοητό αυτό που έλεγα, Πρόεδρε. Μιλώ για τον επαναπατρισμό των παιδιών ξένων μαχητών στη Συρία και στο Ιράκ και των μητέρων τους. Είχαμε λάβει πολύ σαφή θέση το Μάιο Ακόμα πιο ανισχυτική είναι η κατάσταση σήμερα μετά την ε, τουρκική επίθεση. Έχουμε ήδη χάσει τα ίχνη ορισμένων παιδιών και συζύγων μαχητών. Ε, είναι θέμα και ασφαλείας αλλά και ανθρωπιστικό. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια ανάληψη δράσεως από τα κράτη-μέλη που ενέχονται και να υπάρχει ένα ε, συντονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση. Εσείς τι θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει επιγόντω για την κατάσταση στη Συρία. Επίσης, πώς βρίσκεται την πρόταση κάποιων κρατών μελών να συστήσουν ένα δικαστήριο ad hoc για να δικάζουν τους ε, μαχητές αυτούς. Πρόεδρος, ο κύριος Μάρκατ. Ναι, ευχαριστώ. Δύο ερωτήματα. Αφενός, μιλάμε πολύ για την Κεντρική Μεσόγεια και για την κατάσταση που επικρατεί εκεί, κάτι που μας απασχόλησε και με αφορμή το ψήφισμα. Ε, υπάρχει πάντοτε αυτό το pull factor effect που συζητούμε, δηλαδή το ότι η βοήθεια που παρέχεται σε μετανάστες στη Μεσόγειο στην πραγματικότητα δεν βοηθά. Εγώ δεν την κατανοώ πολύ αυτή τη συλλογιστική. Οι προτάσει που γίνονται είναι αφενός να ε, απελάβνονται οι άνθρωποι αυτοί στην Λιβύη ή να μην διασώνονται αυτοί. Αυτό, να μην διασώζονται. Αυτό βεβαίως ε, είναι αδιανόητο. αν δει κανεί το χάρτη και τα πλοία που υπάρχουν από μη κυβερνητικέ οργανώσει στην Μεσόγειο, ε, το ερώτημα είναι ε, επιτρέπεται να επιστρέφονται αυτοί οι άνθρωποι στη Λιβύη. Δεν επιτρέπεται κανείς ε, να διασώζει ανθρώπους που κανονικά υποχρεούνται και με βάση το, το δίκαιο της θάλασσας να το, να το πράττει. Είναι λίγο το ερώτημά μου. Δεύτερο ερώτημα. Η Μάλτα έχει κατηγορηθεί ότι καθυστερεί σκοπίμως ε, τις ε, επιχειρήσεις διάσωσης. Εσείς τι γνωρίζετε όταν υπάρχει πληροφορία ότι υπάρχουν άνθρωποι στη θάλασσα, στη θάλασσα κινούνται άμεσα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να διασωθούν. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. λίγο με Διana Ρίβα από την ε, ομάδα των Πρασίνων ε, και επίσης είμαι σύζυγο του Ραούλ Ρομέδα ε, ο οποίος επί 10 χρόνια ήταν ευρωβουλευτή και μέλο τούτη τη Επιτροπής. Ο Ραούλ Ρομέδα καταδικάστηκε σε 12 χρόνια εγκλισμό ε, την προηγούμενη εβδομάδα για λόγο του ότι οργάνωσε ένα ε, δημοψήφισμα. Γνωρίζετε την κατάσταση στην Καταλωνία, θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό. Η βαριά, η σκληρή ποινή κατά των ε, Καταλανών υπευθύνων για το δημοψήφισμα καταδικάζει την ελευθερία σκέψης και την δημοκρατία. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες είδαμε και αστυνομική η βία που μας αφήνει άφωνους. Ε, οι Ισπανικές αρχές σε συνεργασία με τις καταλανικές ε, αρχές ε, διαρκώς υποδαβλίζουν μία όλο και πιο μεγάλη πολιτική διαφορά. Εγώ θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι ευρωπαϊκό, όχι μόνο ισπανικό και καταλανικό. Και για να σας πω ότι έχουμε 7 ανθρώπους σε φυλακές της Μαδρίτης καταδικασμένους ε, για, τη, για τρομοκρατία, ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει υπάρξει τρομοκρατία ε, στην Καταλωνία. Επίσης υπάρχει ανακριτικό μυστικό και δεν γνωρίζουμε ε, καθόλου όλα τα στοιχεία. Έχουμε 28 κρατούμενους από τις τελευταίες tenido daños διαμαρτυρίες στην ε, Βαρκελόνη, 60 δημοσιογράφου ε, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα και δεν μπορούν να γράψουν αυτά που θέλουν. Εμείς θέλουμε να σταματήσει πια αυτή η κατάσταση στην Καταλωνία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρίβα. Η κυρία Νταλή έχει ζητήσει το λόγο και η κυρία Κέλλερ επίσης. Ε, θα σας δώσω τον λόγο. Δεν είχα ζητήσει τον λόγο, όμως θέλω να πω στην αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, Επίτροπο θα, θα μιλήσω, θα μιλήσω κι εγώ. Αυτό σας λέω, λέει ο Πρόεδρος. Ε, θέλω να ε, μιλήσω στα Ισπανικά ε, για να σας πω ότι θα σεβαστώ όλους όσοι θέλουν να μιλήσουν και σας παρακαλώ να σεβαστείτε και το δικό μου δικαίωμα να μιλήσω. Απλώς σε καμία περίπτωση δεν ε, ε, έχει υπάρξει ποινική ε, δίωξη ή καταδίκη για λόγους ελευθερίας έκφρασης και δημοκρατίας. Πρόκειται εδώ για μια ποινική καταδίκη μετά από κατηγορίες για παράνομο δημοψήφισμα. Παρατηρήσει εκτός μικροφώνου δεν ακούν οι διερμηνείς δυστυχώς. Διαμαρτυρίες από την αίθουσα. Πρόεδρος. Κοιτάξτε, ε, όλοι παίρνουν το λόγο εν πλήρη ελευθερία, όλοι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα του να μιλούν και να ακούγεται ο λόγος τους. Εγώ απλώς ε, λέω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύτηκε ε, το δικαίωμα έκφρασης ή διαδήλωσης. Εδώ μιλάμε για ποινικέ ε, αποφάσεις, μετά από ποινικέ διαδικασίες ε, δηλαδή, ε, που έχουν βασιστεί στο ποινικό κώδικα μιας δημοκρατίας, μιας χώρας τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ήθελα να πω. Διαδικαστικό παρακαλώ. Εσείς ε, είστε πρόεδρος ε, τη επιτροπή, ε, Πρέπει να δώσετε σε όλους την δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήματα ή στην Επίτροπο. Όμως εδώ μετά από μια συγκεκριμένη ερώτηση λέτε ότι έχετε το δικαίωμα να παρέμβετε για να πείτε αυτά που λέει η κυρία δεν είναι σωστά. Δεν είναι όμως αυτή η θέση σας ως πρόεδρος και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να το ξανακάνετε. Πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Εγώ αισθάνθηκα υποχρέωση να το πω ε, γιατί εδώ μιλάμε, απευθυνόμαστε ε, εις την Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις δίνουμε στοιχεία τα οποία δεν είναι σωστά, δεν είναι αληθή και επομένως ε, πραγματικά είμαι υποχρεωμένος να ξεκαθαρίσω τα πράγματα σε σχέση με την ποινή την οποία αποφάσισε ένα ποινικό δικαστήριο βάσει του ποινικού κώδικα της Ισπανίας. Η ελευθερία του συναθρίζεστε, η ελευθερία του, της ε, διαμαρτυρίας, της διαδήλωσης και η ελευθερία έκφρασης ε, διασφαλίζονται στο Σύνταγμα της ε, Ισπανίας εδώ και 40 χρόνια πλέον. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία τέτοια αναφορά και δεν υπήρξε καμία ποινικοποίηση αυτών των στοιχείων. Επομένως, τα πραγματικά περιστατικά είναι διαφορετικά. Τα πραγματικά περιστατικά τα οποία ε, ε, αποτέλεσαν βάση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ε, δεν σχετίζονται με την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία προστατεύονται. Πρέπει, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Και εσείς για διαδικαστικό θέλετε. Πρόεδρε, θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά της συνεδρίασης ότι κάνετε κατάχρηση της θέσης σας προκειμένου να εισαγάγετε το θέμα έτσι όπως θέλετε εσείς στη συζήτηση. Μιλούν και οι, δύο, και οι ομιλητές ταυτόχρονα, και ο πρόεδρος και το μέλος. Αναγκάστηκα, λέει ο πρόεδρος. Όχι, έχετε κάνει κατάχρηση, πρόεδρε, και να μπει στα πρακτικά. Ζητώ. Ο πρόεδρος, πρέπει να ολοκληρώσουμε τον ε, γύρο των ομιλητών. Η κυρία Ντέλη. Ε, πρόεδρε, ελπίζω να μπορέσω να μιλήσω χωρίς να με διακόψει κανείς. Ήθελα να μιλήσω για την ελευθερία έκφρασης. Καταρχάς, ε, σχετικά με το θέμα του Τζούλιαν Ασάνς, που ίσως να γνωρίζετε ότι ήταν στο δικαστήριο σήμερα, του αρνήθηκαν ε, να προετοιμάσει την υπεράσπιση του έναντι της πιθανής του έκδοσης, όπου αντιμετωπίζει 170 ε, χρόνια φυλάκιση σωρευτικά είναι η περίπτωση σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς και ήθελα να ξέρω τι κάνετε εσείς ή ποια είναι η θέση σας σχετικά με αυτό. Επίσης, για την θέση στην Καταλωνία θέλω να πω το εξής. Ε, είναι γεγονός ότι έχουμε υπουργούς, εκλεγμένους αντιπροέδρους, οι πολιτιστικούς ηγέτες, οργανώσεις που όλοι πάντοτε ήταν υπέρ του ειρηνικού διαλόγου σε όλες τους τις τοποθετήσεις και έχουν φυλακιστεί 9 έως 13 χρόνια. Υπήρχε λοιπόν ένας κίνδυνος, ε, νομίζω πλήττεται το δικαίωμά τους να λάβουν δίκαιη ακροαματική διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου. Υπάρχουν ε, χιλιάδες ανθρώπων στο δρόμο στην Καταλωνία. Η αστυνομία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη μαζική αντίδραση του πληθυσμού. Εγώ έχω φίλους στην πόλη αυτή, έχω δει σκηνές βίντεο, είναι σαν εμπόλεμη ζώνη. αστυνομική με ειδικό εξοπλισμό μάχης εγώ ντρέπομαι να μιλούμε σε φόρουμ σαν αυτό εδώ, το σημερινό, για ανθρώπινα δικαιώματα και να έχουμε τέτοια φαινόμενα στις χώρες μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε να μιλούμε διαρκώς, συνεχώς όλοι και θέλω να ξέρω τι κάνετε εσείς. Η κυρία Κέλλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο που βρήκε το χρόνο Ίσως χρησιμοποιήσει αυτή τη μικρή δίωδο, το τούνελ που ενώνει τα κτηριά μας εδώ με το Συμβούλιο της Ευρώπης που είναι, συμβολίζει έναν σύνδεσμο αλλά βέβαια δεν μιλώ αντικειμενικά. Ε, εγώ είμαι από το Στρασβούργο και μ' αρέσει αυτή η κυκλοφορία, η ελεύθερη κυκλοφορία προς όλες τις κατευθύνσεις, ώστε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρώπης. Και σε κοινά θέματα που εξετάζουμε εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και εσείς στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εμπίπτουν απολύτως στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας. Ήθελα λοιπόν τρία σημεία να σας ε, διαβιβάσω. Ε, αναφερθήκατε στην απόφαση της Μάλτας και εκφράσατε τη λύπη σας, ε, όπως και εμείς, που δεν συμμετέχουν περισσότερα μέλη. Τι πρωτοβουλίες θα μπορούσαμε να αναλάβουμε. Εσείς ως Συμβουλίο της Ευρώπης, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ενθαρρύνουμε και άλλα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν. Ε, υπογραμμίσατε και δεν είμαι σίγουροι ότι κατάλαβα απόλυτα καλά. Υπογραμμίσατε πάντω τη σημασία τη συνεργασία με τρίτε χώρε ή στα πλαίσια τη μετανάστευση. Ο κύριο Μπορέλ στην ακροματική του διαδικασία και αυτός αναφέρθηκε σε αυτή τη συνεργασία. Εσείς τι είναι το αρνητικό που βλέπετε εκεί, μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο. Και ένα ευαίσθητο ερώτημα αυτό το τελευταίο που θα σας κάνω. Λεπτό ερώτημα. Εσείς γνωρίζετε τι συμβαίνει στα στρατόπεδα των προσφύγων από τη Συρία που βρίσκονται στην Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δυστυχώς έχει πολύ περιορισμένε δυνατότητε να γνωρίζει τι σημαίνει εκεί. Εσείς μήπως γνωρίζετε κάπω περισσότερα πράγματα. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Κάποιο άλλο μέλος, λέει ο Πρόεδρος. Όχι. Κανένα άλλο μέλος. Ο κύριος Μπουσαντέ. Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, ήμουν στην Ολομέλεια και μόλις γύρισα στην αίθουσα άκουσα να αναφέρονται διάφοροι στην πόλη μου, στην Βαρκελόνη. Γίνεται λοιπόν προπαγάνδα εδώ πέρα. Fake news ακούμε από εκείνους που είναι υπέρ των, της, ε, του κινήματος ανεξαρτησίας είχαμε πράξεις βίας, και ένα κτίριο από αυτούς τους διαδηλωτές υπέρ της αναξαρτησίας της Καταλωνίας και ε, τέθηκαν ζωές και μικρών παιδιών σε κίνδυνο. Εδώ μιλούμε για ανθρώπους, άτομα που έχουν καταδικαστεί με ποινικέ αποφάσεις και έχουν, έχουν καταδικαστεί για στασιασμό από δικαστήριο 500 ετών ιστορίας, νομολογίας, συντάγματος με διατάξεις. Δεν, μπορούν, δεν μπορείτε να κάνετε λοιπόν δηλώσεις ε, του τύπου σαν αυτές που ακούμε εδώ στην αίθουσα αυτήν. Είχαμε αποφάσεις με κάθε νομιμότητα και σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα για την πανέμορφη πόλη της Βαρκελόνης και για την όμορφη χώρα μας όταν υφίσταται αυτή η πανέμορφη πόλη οι επιθέσεις, πυρκαγιές, βίαιες επιθέσεις κίνδυνος για τους πολίτες, για τους κατοίκους της πόλης κίνδυνος για εκπρόσωπους, για εκπρόσωπους τύπου, για δημοσιογράφους από ορδές ε, διαδηλωτών εν εξάλλου. Επομένως, αν θέλετε να τοποθετήσετε για το θέμα, ε, να σέβεστε σας παρακαλώ την, την ε, αρμοδιότητα του Ισπανικού κράτους να χειρίζεται το θέμα αυτό το εσωτερικό και τις καταστάσεις όπως έχουν στο πεδίο, στο έδαφος. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, ακούσαμε τα μέλη, ακούσαμε τις ερωτήσεις. Τώρα, Επίτροπε, σας παρακαλώ Ομοδοποιήστε βεβαίω όπως θέλετε τις διάφορες ερωτήσεις και παρατηρήσεις που ακούστηκαν προκειμένου να μπορέσετε αν θέλετε να θίξετε όλα αυτά τα κεφάλαια. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλους για τις πολύ σημαντικές ερωτήσεις που μου απευθύνατε, τα πολύ σημαντικά σημεία, θέματα που θέσατε θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα και θα προσπαθήσω να ε, απαντήσω ε, κατά ομάδες. Εν τούτης είναι πολύ σημαντικό και θέλω να σας το πω για να μην το ξεχάσω ότι μπορείτε πάντοτε να ε, απευθύνετε τέτοιου είδους ερωτήματα ε, στο επιτελείο μου. Θεωρώ ότι Πάρα πολλά από αυτά τα ζητήματα θα μας απασχολήσουν και στις μελλοντικέ μας συζητήσεις. Και συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπε η κυρία Κέλλερ, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις γέφυρες που έχουμε χτίσει για να μπορέσουμε να επιφέρουμε απτά αποτελέσματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρώτα απ' όλα, πολλοί από εσά αναφερθήκατε στην Τουρκία για διάφορους λόγους. Μετανάστευση, την τρέχουσα συγκυρία αλλά και την ελευθερία έκφρασης. Η εντολή μου είναι αρκετά περιορισμένη. Εγώ είμαι υπεύθυνη για 47 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν έχω εντολή να παρεμβαίνω ε, ή να παρέμβω στην Συρία. Υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Ωστόσο βεβαίως παρακολουθώ την κατάσταση όχι μόνο την κατάσταση στη Συρία, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, προκειμένου να μπορώ να διαμορφώνω μια συνολικότερη εικόνα και να μπορώ να βλέπω πώ επηρεάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, είτε των Ευρωπαίων πολιτών, είτε ε, των ανθρώπων που βρίσκονται σε ε, εμπόλεμε ζώνε. Παρακολουθώ λοιπόν την κατάσταση στην, στην Συρία και στην Τουρκία όσον αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης. Και νομίζω ότι αυτό το θέμα θα παραμείνει πολύ ψηλά στην ατζέντα μου και σκοπεύω να επανέλθω σε επαφές ε, με τις τουρκικές αρχές για το ζήτημα αυτό. Εγώ στη διάρκεια της ε, μέχρι τώρα θητείας μου έχω επισκεφτεί ήδη δύο φορές την Τουρκία, ωστόσο προτεραιότητα είχαν άλλα καυτά θέματα τα οποία επίσης βρίσκονται στην ατζέντα μου, όπως είναι η κατάσταση ε, των ε, δημοσιογράφων και των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και το ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης που επηρεάζει συνολικά την κοινωνία των πολιτών. Θα δημοσιεύσω έκθεση ε, για την Τουρκία τον Ιανουάριο του 2020 και εκεί θα ε, αναφέρομαι ρητός στο ζήτημα των ε, δημοσιογράφων, των υπερασπιστών των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Είχα επίσης την ευκαιρία να έχω πρόσβαση σε φυλακές στην Τουρκία. κατάφερα και συναντήθηκα με τον Άχμετ Άουταν, με τον Όσναρ Κάβαλα και έναν δικηγόρο προκειμένου να διαπιστώσω η διεισόμαση, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, που κρατούνται και βεβαίως θα ε, αναφερθώ και σε αυτά στην έκθεσή μου. Βεβαίως λαμβάνω υπόψη μου και την κατάσταση στην Συρία και πιθανά ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση και που ενδεχομένως επηρεάσουν ε, ανθρώπους που ε, βρίσκονται εκεί. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να πω το οτιδήποτε, διότι δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες. Βεβαίως βρισκόμαστε σε επαφή ε, και σε συζητήσεις με μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να, να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και να προετοιμάσουμε μια ενδεχόμενη παρέμβαση αλλά σας ξαναυπενθυμίζω αυτόν τον περιορισμό το, της εντολής μου. Εγώ έχω αρμοδιότητα και ευθύνη για τα μέλη του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Όσον αφορά την ε, Μάλτα και την ε, Δάφνη, πολλοί από σας θέσατε το ζήτημα αυτό μια υπόθεση η οποία συγκλώνησε την Ευρώπη και όχι μόνο την Ευρώπη. Εγώ δεν θα επισέλθω σε εκτιμήσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις, τις συνέπειες της έρευνας που έχει διεξαχθεί, ούτε στο πώς ε, έχει χειριστεί το ζήτημα η μαλτέζικη κυβέρνηση. Νομίζω ότι ήμουν σαφής και στην ανακοίνωσή μου, αλλά και στην επιστολή που απίφθηνα ε, στον Πρωθυπουργό κύριο Μουσκάτ και του ζήτησα να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει η μετά θάνατον κατασυγκοφάντηση της δημοσιογράφου αυτή, ε, αυτής. Υπάρχουν, λοιπόν, ένα, υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα ατιμορρησίας καθώς και άλλα ζητήματα που μπορεί κανείς να θέσει όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και ξέρετε ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει ξεκινήσει και μια ε, ειδική ε, εξεταστική επιτροπή για το ζήτημα. Και υπάρχουν και πάρα πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες διασφαλίζουν ότι το θέμα δεν θα ξεχαστεί. Εγώ από την πλευρά μου θα συνεχίσω βεβαίω τη συνεργασία μου και με αυτέ τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και με όλου του φορεί, αλλά και βεβαίω και με την κυβέρνηση τη Μάλτα, προκειμένου να διελευκανθεί η σκοτεινή αυτή η υπόθεση και για να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Γιατί αυτό, όπως είπα και στην ε, δήλωσή μου, το χρωστάμε στη Δάφνη, στην οικογένειά τη και σε όλου του δημοσιογράφου σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλοί αναφερθήκατε επίση στην ε, πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα της μετανάστευσης και στο γεγονός ότι 7 ή μόνο 12 κατά άλλε πηγές συμφώνησαν να συνεργαστούν και προσπάθησα με την δήλωση την οποία εξέδωσα να έρθω σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε ζητήματα μετανάστευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πολύ νωρίς ε, να πω μια οριστική γνώμη, όμως σαφές είναι το εξής. Ό,τι γίνει θα πρέπει να γίνει με τρόπο συμβατό με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που είπα και εισηγητικά και που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι είναι πολύ ντροπιαστική η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη όταν μιλάμε για αλληλεγγύη όλων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον ε, δίκαιο επιμερισμό των βαρών ε, που αυτή τη στιγμή έχουν ε, κατά κύριο λόγο επομιστεί συγκεκριμένες χώρες. Και επανέρχομαι εδώ στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα πραγματικά αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα υποδέχεται τεράστιο αριθμό ανθρώπων και δεν έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί ε, ένα, μια τόσο μεγάλη ροή μεταναστών και δυστυχώς δεν έχει δεχτεί ε, τον, ε, την αλληλεγγύη των άλλων κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και εσείς επίσης αναφερθήκατε και στο, στο, στην στο αίτημά μου να κλείσει το στρατόπεδο στην ε, Βοσνία Ερζαγωμίνη. Για μένα, ξέρετε, είναι και συναισθηματικό το ζήτημα. Θεωρώ ότι είναι ντροπή. Ο λαός της Βοσνίας Ερζεγοβίνης να μην επιδεικνύει αλληλεγγύη απέναντι στους πρόσφυγες που δεν επιδεικνύει την απαραίτητη συμπόνια που θα περίμενε κανείς γιατί μόλις πριν από 20 χρόνια βρεθήκαμε κι εμείς οι ίδιοι οι Βόσνοι σε μια παρόμοια κατάσταση και αναζητούσαμε χώρο ασφαλή όπου θα μπορούσαμε να, να ζήσουμε. Τώρα φαίνεται δυστυχώς ότι η αλληλεγγύη και οι άλλες αρχές που μας διακρίνουν ως ανθρώπους ε, φαίνεται να εγκαταλείπονται. Δεν έχει σημασία όμως, η φωνή μας πρέπει να ε, ακουστεί. Βεβαίως δεν μπορώ μόνη μου ε, με την υπηρεσία μου να λύσω το τεράστιο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μετανάστευσης. Λέω όμως ότι θα πρέπει πραγματικά να ενώσουμε τις φωνές μας για να μπορέσουμε να επιφέρουμε αλλαγές και να υπάρξει μια πραγματική μεταστροφή. Και αυτό είναι και ένα σημαντικό καθήκον της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δικό σας ε, καθήκον ως Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ε επίσης είναι να κατευθυνθείτε να προχωρήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά όχι μόνο εσεί, είναι και η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για του πρόσφυγε, καθώ και πολλοί άλλοι φορεί που συμβάλλουν στο να γίνει πιο διαχειρίσιμο το πρόβλημα. Αυτό όμω που λείπει είναι η πολιτική βούληση. Γι' αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Εδώ, ε, σε πολλά θεσμικά όργανα στην Ευρώπη, δυστυχώ. Ε, είναι μια πραγματικότητα και πρέπει με θάρρος να προχωρήσουμε για να ανατρέψουμε, να αναιρέσουμε αυτήν την τροπιαστική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και να επαναφέρουμε ε, και να αποκαταστήσουμε την Ευρώπη ως ε, περιοχή του κόσμου όπου γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά δείγματα περί του αντιθέτου. Ωστόσο υπάρχει ελπίδα, υπάρχουν οι αξίες μας και αυτές πρέπει να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά όπω είπα, πολύ συχνά τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται μόνο στα χαρτιά και όχι στην πράξη. Αυτό που εγώ μπορώ να κάνω ω επίτροπο είναι το εξή. Μπορώ να χρησιμοποιήσω διάφορα εργαλεία. Καταρχά, μπορώ να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου, που είναι και το πιο ισχυρό εργαλείο που έχω στα χέρια μου. Αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω και να αξιοποιήσω και άλλου μηχανισμού που έχω στη διάθεσή μου. Από παρεμβάσει ε, τρίτων έω επισκέψει σε χώρε, την έκδοση δηλώσεων και αυτό το κάνω συχνά, διαρκώς μάλλον, οι παρεμβάσεις ε, σε ε, διάφορα φόρα ε, είναι κάτι που το αξιοποιώ ως εργαλείο διαρκώς. Υπάρχει και ο κανόνας 9, τον οποίο ενέκριναν οι υπουργοί του Συμβουλίου της Ευρώπης και με την, τον οποίο δίνονται ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες στον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Βεβαίως θα πρέπει πολύ προσεκτικά να ε, διαλέξω ποιες είναι οι υποθέσεις ε, εκείνες που κατά προτεραιότητα θα πρέπει να ε, τεθούν υπό επεξεργασία προκειμένου να ασκηθεί πίεση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. όμω θα σα ενημερώσω ε, μόλις ληφθούν σχετικές αποφάσεις. Έχω ήδη λάβει τέτοιες αποφάσεις για το ζήτημα της μετανάστευσης, των υπερασπιστών, των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφων, των ΑΜΕΑ, καθώς και ε, τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταναστών. Προσπαθώ πραγματικά τη θέση μου να την αξιοποιήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να συμβάλλω θετικά στην επίλυση των πλέον προβληματικών καταστάσεων. Εγώ παρακολούθησα με πολύ προσοχή τις, ε, τις ακροάσεις των ορισθέντων επιτρόπων και η κυρία Κέλλερ αναφέρθηκε και στον κύριο Μπορέλ και τις απόψεις που εξέφρασε και γνωρίζω ότι Οι τρίτε χώρε αναφέρθηκαν με διάφορε αφορμές. Για μένα το ερώτημα δεν είναι αν τα κράτη-μέλη συνεργάζονται με τρίτες χώρες, αλλά το αν θα το κάνουν με διαφανή τρόπο που θα εξασφαλίσει τη λογοδοσία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι το βασικότερο ζήτημα. Φυσικά, ε, συνεργασία δεν, δεν, δεν, δεν θα πω εγώ σε κανέναν επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αν θα προχωρήσουν σε συνεργασία ή όχι. Όμως, ο τρόπος με τον οποίο θα διαμορφωθεί αυτή η συνεργασία και το αν θα γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτό είναι ένα ζήτημα που με, που απασχολεί και όπου θα παρεμβαίνω. Αναφερθήκατε και στο ζήτημα της, ε, του, των απόψεων του Πάπα για τη μετανάστευση. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη και να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ε, θεωρώ από αυτή την άποψη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θρησκευτικοί ηγέτες να μιλούν εξ ονόματος των ανθρώπων και να θέτουν ε, ανθρώπινα δικαιώματα, ε, ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τα αναδεικνύουν. Το, το λόγος μίσους επίσης ε, αναφέρθηκε. Ε, επ' αυτού είναι αμφιλεγόμενες οι απόψεις. Γιατί ναι, εγώ θέλω την ελευθερία έκφρασης. Ε, θέλω την αποποινικοποίηση, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνουν περισσότερα από τα κράτη-μέλη, γιατί υπάρχουν ακόμα χώρες-μέλη που δεν, ε, ε, δεν έχουν αυτήν την απαραίτητη αποποινικοποίηση. Φαντάζομαι επίσης ότι δεν είναι δυνατόν τέτοιου είδους περιορισμοί να δίνουν την δυνατότητα να σταματήσουμε ας πούμε απόψεις ή να αποκλείσουμε απόψεις ε, που δεν μας ενδιαφέρουν. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να γίνουν χιδαίοι, άνθρωποι που θέλουν ε, να γίνουν προκλητικοί. Ε, δεν είναι δυνατόν να πέφτουμε στο παιχνίδι αυτών των ανθρώπων. Βεβαίω, ο, ο λόγος δεν εμπίπτει στο δικαίωμα ελεύθερης έκφραση. Αυτό είναι σαφές και από αυτού οπωσδήποτε θα συνεχίσω να εκφράζω την άποψη άποψή μου και μάλιστα πολύ φωναχτά. Η Ρωσία αναφέρθηκε επίσης. Ε, πανέρχομαι στην ε, ε, κοινοβουλευτική συνέλευση. Εγώ είμαι επίτροπος ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ξέρω ποιος είναι ο ρόλος μου ε, και ξέρετε πολύ μεταξύ ημών ότι δεν φοβάμαι καθόλου να πω την άποψή μου. Η Ρωσία όμως είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και οπωσδήποτε θα επισκεφθώ τη Ρωσία όσον ούπο τον Απρίλιο συγκεκριμένα. Αυτό που θέλω να κάνω ε, είναι πραγματικά να δουλέψω για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσική Ομοσπονδία. Θέλω να πάω στο Βόρειο Κάφκασο, θέλω να πάω σε όλες αυτές τις ε, ε, περιφέρειες τις οποίες κανείς δεν επισκέφτηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από το 2014 και μετά κανένας Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν επισκέφτηκε αυτές τις περιοχές και οπωσδήποτε θέλω να ξεκινήσω με τις ρωσικές αρχές συζητήσεις έτσι ώστε να συζητήσουμε τα πολλά ζητήματα προβληματισμού Όσον αφορά το θέμα της Κρυμαίας, πολύ σημαντικό Βεβαίως προτίθεμαι ε, να ε, επισκεφτώ την Κρυμαία αλλά και άλλες ε, λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Όλοι όσοι ζουν υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να έχουν το δικαίωμα της προστασίας. Τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει οπωσδήποτε να δεσμεύονται κατά την έννοια αυτή. Και αυτό είναι και δική μου προτεραιότητα. Βεβαίως οι ευαισθησίες είναι πολλές, είναι γνωστές, το πολιτικό περιβάλλον επίσης είναι γνωστό. Γνωρίζουμε ότι αυτό καθόλου εύκολη δουλειά δεν είναι. Το, με ρωτάτε αν θα συζητήσω το θέμα με τις Ουκρανικές αρχές. Φυσικά είναι αυτονόητο. Εάν επισκεφθώ την ε, Κρυμαία όλα θα γίνουν ε, σύμφωνα με το γράμμα του διεθνούς δικαίου ε, και της νομοθεσίας. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις ε, ε, θα πάω στην Κρυμαία και είναι σημαντικό να επισκεφθώ την Κρεμία. Προς ώρες δεν μπορώ να σας πω πότε θα γίνει αυτή η επίσκεψη, όμως ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι προσπαθώ να έρθω σε επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και προτίθεμαι πολύ σύντομα να επισκεφθώ και το Κίεβο πριν το τέλος του 19 έτσι ώστε να έχουμε συζητήσεις και από αυτού μεταξύ και άλλων πολλών θεμάτων ε, θα πάω και μετά από την επιστροφή μου ε, βεβαίως με μεγάλη χαρά να ξαναέρθω στην Επιτροπή σας για να συζητήσουμε γι' αυτό. Προς ώρας πάντως δεν μπορώ να σας πω τίποτε περισσότερο καθότι οι συζητήσεις δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Uh, uh, Πολωνία, νομίζω ότι υπήρξα σαφής στη διάρκεια της συζητήσεως ε, επί του θέματος αυτού. Η ημερομηνία, αν δεν ε, σφάλω, τότε δηλαδή που έκανα μία δήλωση, δεν θυμάμαι ακριβώς ε, Είναι πολλές ερωτήσεις. Ο Πρόεδρος ζητά από την κυρία Επίτροπο να συντομεύσει όσον αφορά την Καταλωνία. Δεν θέλω να μπω πολύ στην συζήτηση αυτή. Εγώ έκανα μία δήλωση, την οποία θα σας ζητήσω να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μου. Έχω βεβαίως επαφές και είχα σε ε, πολλές περιπτώσεις την ευκαιρία να συναντήσω Ισπανούς πολιτικούς με τους οποίους έθιξα αυτό το ζήτημα. Δεν πρόκειται για νέο πρόβλημα. Η Ισπανία ως ε, χώρα ε, είχε πρόβλημα όσον αφορά την ε, αρχή του συναθρίζεστε ε, και το είχε καταδείξει και ο προκάτοχός μου. Προτεθήμαι λοιπόν να συζητήσω με τις Ισπανικές Αρχές για τα θέματα αυτά. Βεβαίως αυτό που βλέπω τώρα είναι ακριβώς το θέμα της ελευθερίας συνάθρησης, γιατί αυτό είναι καυτό θέμα. Τα παιδιά στην Συρία, πολύ σημαντικό είναι ένα ζήτημα το οποίο ήδη έχω θίξει. Το έχουμε συζητήσει επίσης και με άλλους διεθνείς οργανισμούς, κυρίως με τα Ηνωμένα Έθνη. Γνωρίζω δε τις διάφορες προτάσεις οι οποίες έχουν προκύψει. Για την ώρα πάντως το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι παρακολουθώ το θέμα με μεγάλη προσοχή κυρίως όσον αφορά τα παιδιά. Θα μπορούσα να μιλάω επί ώρες, ε, αλλά ξέρω ότι δεν έχω όλο το χρόνο που θα ήθελα στη διάθεσή μου. Γι' αυτό θα πρέπει να σταματήσω. Ε, αν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μου, στείλτε μου ένα ε, email και ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα ξανασυναντηθούμε διαζώσεις. Ε, αυτό και η σημερινή μας συζήτηση άλλωστε καταδεικνύει πόσα είναι τα ζητήματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, θέλουμε να συζητήσουμε και πολλά ε, επί των οποίων μπορούμε να συνεργαστούμε. Σας ευχαριστώ και εμείς σας ευχαριστούμε λέει ο Λοιπόν, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον προκάτοχό σας. Έχετε ακόμα αρκετό καιρό στην δική σας θητεία να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε την συνεργασία. Βεβαίως και τα μέλη είναι ελεύθερα πάντοτε να επικοινωνούν μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αλλά έχουμε ακόμα δύο σημεία για την σημερινή μας συνεδρίαση, οπότε θα σας ευχαριστήσω εδώ θερμά και θα καλέσω τους συναδέλφους να πάμε απευθείας στο επόμενο σημείο, που είναι η ανταλλαγή σχετικά με την ε, Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και το σύστημα ΦΑΝΤΟ για την ε, κοινή δράση 19.700. Η κυρία Μετσόλα έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχουμε λάβει 73 τροπολογίες από όλο το πολιτικό φάσμα. Κάτι λέει ο πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Να ακούσουμε την συγγήτριά μας, την κυρία Μετσόλα, για το φάντο. Ναι, λοιπόν, έλεγα τροπολογίες από το σύνολο του πολιτικού φάσματος για την πρόταση Φαντό, μαζί και με, αυτή, και με αυτές που εγώ είχα υποβάλει στο σχέδιο έκθεσης. Ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα όλους τους συναδέλφους για την συμμετοχή, την συζήτηση, εν ώψη των διαθεσμικών διαπραγματεύσεων με Συμβούλιο και Επιτροπή αργότερα φέτος και προκειμένου να έχουμε συνέχεια με το παρόν σύστημα φάντο, μιλούμε για αυθεντικά ή γνήσια έγγραφα και διευκρινίζουμε τι εννοούμε. Μιλούμε για τη διατήρηση του πεδίου εφαρμογή όπω και στην αρχική πρόταση, αλλά με διαφορετικέ υποχρεώσει για το τι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει. Το, οι SD διατηρούν το δικαίωμα πλαστοποιημένων ταξιδιωτικών εγγράφων ή αδειών παραμονής ή αδειών οδήγησης ή αδειών κυκλοφορίας. Αλλά με τις ίδιες τροπολογίες το φάντο μπορεί να συμπεριλαμβάνει και άλλα επίσημα έγγραφα σχετικά με ταξιδιωτικά ε, έγγραφα, έγγραφα ταυτοποίησης ή άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας είναι θέματα δομή του φάντο σχετικά με το ποιο θα έχει πρόσβαση. Υπό του πράσινου, έχουμε μια διάκριση μεταξύ των τρίτων μερών, τρίτων χωρών δηλαδή και αερομεταφορέων. Αλλού δεν έχει γίνει αυτή η διάκριση, αυτή η διαφοροποίηση. Υπάρχει επίση υπάρχει μια ρήτρα ΜΕΙ σχετικά με την επικράτεια τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών. Είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά, διαπραγματευόμενοι τι συμβαστικέ τροπολογίες. Επίσης περιμέναμε να λάβουμε μεγάλο αριθμό για την επεξεργασία των δεδομένων. Τα περισσότερα μέλη έχουν αντίστοιχες απόψεις από αυτού, σύμφωνα δηλαδή με τις ε, προτάσεις τροπολογίες που έχουμε λάβει. Είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να βρούμε μια πολιτική συμφωνία που θα λαμβάνει υπόψη της όλα, όλες τις οπτικές γωνίες. Και άλλες τροπολογίες που υπευλήθησαν για την ενίσχυση της συνεργασίας με τον Frontex και τον EU Lisa. Αυτό το πρώτο είναι το Renew. Όπως και το, τη δυνατότητα της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου να διαβιβάζει τα δεδομένα του υφιστάμενου φάντου, φάντο στο νέο σύστημα χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών. Αυτά συνοπτικά. Έχουμε άλλη μια συνάντηση ε, των σκιωδών για αύριο εγώ περιμένω με ενδιαφέρον τη συνέχιση τη δουλειά αυτή με του υπόλοιπου σιώδεις. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ευρύτατη στήριξη των περισσότερων πολιτικών ομάδων. Ε, ευχαριστούμε κυρία Μετσόλα. σας ακούσουμε τον, τους Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ε, με ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή συνεργασία και την πολύ καλή δουλειά. Ένα-δύο θεματάκια έχουν ήδη επιληθεί. Ε, από αυτά που εκκρεμούν ήθελα να αναφερθώ στα πιο σημαντικά για εμένα. Καταρχάς έχουμε το θέμα των προσωπικών δομένων στο Φάντο. Με τους κοιόδης και από τις συναντήσεις με Συμβούλιο και Επιτροπή λάβαμε λεπτομερή εξήγηση για ποιον λόγο κάποια προσωπικά δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται στο Φάντο. Ότι δηλαδή οι αναπαραστάσεις, μάλλον οι εικόνες προσώπου ε, είναι τέτοιες στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να αποφύγουν και την απεικόνηση, δηλαδή την φωτογραφία του προσώπου. Εκεί δηλαδή όπου τα στοιχεία της ασφαλείας του εγγράφου δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν από την απεικόνηση. Αλλά αυτή η διαφοροποίηση φαίνεται να είναι ο ασφαλέστερος τρόπος ώστε να υπάρχει περιορισμό στην δυνατότητα αποθήκευση προσωπικών δεδομένων και για το υπόλοιπο της πρότασης που θα διευκολυνθεί πάρα πολύ εάν δεχθούμε αυτή τη διάκριση. Σας ευχαρίστησα ήδη και εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου για την απόπειρά σας να περιορίσει την διατύπωση του κειμένου που αναφέρεται στην αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων, αλλά εξακολουθώ να συστήνω στους σκιώδεις και σε εσάς να μην υιοθετήσετε μια ανοιχτή προσέγγιση λευκής επιταγής για τα προσωπικά δεδομένα και την αποθήκευσή του στο φάντο, που πραγματικά θα πρέπει να τα χρειάζεται το σύστημα για λόγους ασφαλείας και αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται. Επίσης, σχετικά με τις κατηγορίες των προσώπων. Η ανάληψη μέτρων υπό το φάντο ή στο πλαίσιο του φάντο θα πρέπει να γίνεται μέσω κατεξιοδότηση πράξης. Και χαίρομαι που βλέπω ότι προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά αυτές οι έξι διαφορετικές κατηγορίες αρχών και προσώπων που θα απαιτείται για αυτές πρόσβαση, είναι ασαφής κατά πόσον η πρόσβαση αυτή θα ήταν διακριτή για κάθε κατηγορία. Έχουμε τον αριθμό των κατηγοριών και έχουμε και ένα επίπεδο πρόσβασης που είναι ο ίδιος. Και όλα αυτά είναι λίγο συγκεχημένα. Ε, θα εκτιμούσα λοιπόν να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό, να επιλύσουμε και τα υπόλοιπα εκκρεμή ζητήματα. Um, Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει, για την οργάνωση των συζητήσεων, για τις τροπολογίες, για τον τρόπο με τον οποίο τις έχουμε επεξεργαστεί. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ καλύτερη δουλειά από ό,τι έχουν κάνει η Επιτροπή και το Συμβούλιο, αν δει κανείς το κείμενο που έχουμε ετοιμάσει εμείς σε σχέση με την αρχική πρόταση, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι η πρόοδος είναι προφανής. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να βρούμε σωστές διατυπώσεις προκειμένου Πρώτον, να αποσαφενιστεί το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε με καλύτερο τρόπο να ε, ρυθμίσουμε το ζήτημα της χρήσης των προσωπικών δεδομένων και νομίζω ότι το κείμενο που ε, έχουμε πλέον μπροστά μας είναι ένα καλό κείμενο. Επίσης, χαιρετίζω την προσθήκη, ε, την προσθήκη νέων κατηγοριών εγγράφων στο σύστημα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα έγγραφα βάσης ε, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την αξιοπιστία ταξιδιωτικών εγγράφων ή άλλων εγγράφων που εκδίδονται στη βάση άλλων ε, εγγράφων. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ ε, σημαντικό, μια πολύ σημαντική ένδειξη προόδου. Επίσης, για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ευθύνη των κρατών μελών όσον αφορά την τροφοδοσία πληροφοριών, την κοινοποίηση πληροφοριών, την ε, παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών, την ανάρτηση αυτών των πληροφοριών ε, στο, στα διαδικτυακά συστήματα, στα ηλεκτρονικά συστήματα και χαιρετίζω αυτό στο οποίο έχουμε καταλήξει εμείς. Και τέλος η Γιουλίσα, κάναμε την πρόταση εμείς αυτή, γιατί θεωρούμε ότι με την τεχνική εξέλιξη του κειμένου ε, οι γνώσεις και η εμπειρογνωμοσύνη του Ιουλίσα είναι κάτι που πρέπει να αξιοποιηθεί Υπάρχουν ε, ήδη κάποιες ε, μονάδες ε, στα οποία ο EU Lisa, ο Frontex και άλλοι φορείς πρέπει να συνεργάζονται μάλλον και νομίζουμε ότι πρέπει σε αυτά να συμπεριληφθεί και το σύστημα ΦΑΝΤΟ. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να ξαναευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και ιδίως την εισηγήτρια για όλη τη δουλειά που έχει γίνει. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Μπρικμό. Ευχαριστώ πολύ κυρία εισηγήτρια, ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους που εργάστηκαν επί του θέματος αυτούς και για τις συμβαστικές τροπολογίες. Ε, μας αρέσει ε, αυτή η εκδοχή γιατί είναι ποιοτικό το περιεχόμενο και γιατί ε, ε λαμβάνει υπόψη ε, και το θέμα του περιεχομένου αλλά και το θέμα της πρόσβασης τρίτων ε, μερών όπως αναφέρατε και εσείς. Υπάρχει όμως και ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει καλυφθεί για την ώρα δηλαδή η ευθυγράμμιση του κανονισμού ΦΑΝΤΟ με τον 15-17-25 ε, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων στα αγγλικά, έτσι όπως αναφέρεται στον κανονισμό, λέει δεσμευτικές ε, συμφωνίες, binding and enforceable agreements. Ε, νομίζουμε ότι με αυτήν την με αυτήν την διατύπωση η οποία δεν ε, αναφέρεται στην περίπτωση του Φάντο θα είναι πιο σαφής ο δεσμευτικός χαρακτήρας θα έχουμε όμως τη δυνατότητα να το ξανασύζουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Ταρντίνο. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους συναδέλφους ε, για την εργασία που έγινε. Όπως επανειλημμένα ε, έχω πει και στη διάρκεια της παρουσίασής σας η πρόταση ήταν ένα καλό σημείο εκκίνησης βελτιώσιμο. Δεν έχουμε υποβάλει όμως ε, ε, τροπολογίες. Ε, στην τεχνική συζήτηση για τις συμβαστικές τροπολογίες έγιναν πολλά βήματα προς τα εμπρός όσον αφορά την επαλήθευση και τον έλεγχο. Βέβαια έμειναν και πολλά ζητήματα ανοιχτά για συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο επί των οποίων νομίζω ότι σε γενικές γραμμές μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Ο γενικότερος στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος και η βελτίωση επίσης Τη ε, χρήση προσωπικών και διατήρηση προσωπικών ε, στοιχείων ε, και δεδομένων. Όσον αφορά την επιλογή μεταξύ εφαρμοστικών πράξεων και κατεξουσιοδότηση, νομίζουμε ότι η απόφαση είναι σωστή. Ε, επίσης ε, παραμένουν και κάποια τεχνικά ζητήματα και τα οποία θεωρώ ότι μπορούν να ρυθμιστούν με εφαρμοστικές ε, εκτελεστικές πράξεις όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπουσάντε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι για την εργασία της την οποία θεωρούμε με θετικό πρόσημο. Ωστόσο από αυτές τις πολλές τροπολογίες και και τροποποιήσεις ε, εν τέλει ε, υπάρχει ένα κακό ε, αποτέλεσμα, δηλαδή δεν είναι αποτελεσματικό το σύστημα, γιατί μετά από τόσους ελέγχους και τόσες ε, τελικά πραγματικά δεν είναι αποτελεσματικό. Ενώ αυτό είχαμε πει ήδη από την πρώτη φορά, ότι θέλουμε να είναι αποτελεσματικό το εργαλείο αυτό. Θέλουμε μέσα από κατεξουσιοδότηση πράξης ή e ε, εκτελεστικές ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε λίγο περισσότερο με την θέση του Συμβουλίου που μας φαίνεται πιο λογική. Να λάβουμε υπόψη επίσης ε, το, το, το ίδιο το έγγραφο, γιατί εδώ αναφερόμαστε στο έγγραφο και όχι στην προστασία των δεδομένων, γιατί το θέμα των παραποιημένων εγγράφων ανθρώπων που μπαίνουν και κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και ε, βεβαίως εμείς ε, παρότι δεν συμφωνούμε με όλες τις συμβαστικές τροπολογίες θα προσπαθήσουμε ε, να έχουμε ε, μια επικοδομητική στάση όσον αφορά τώρα αυτήν την διαφοροποίηση όσον αφορά την φωτογραφία που ακολουθεί το έγγραφο. Ε, επαναλαμβάνω και εδώ αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ε, βάζοντας τόσες πολλές δικλίδες και τόσες πολλές ε, προϋποθέσεις, πραγματικά γίνεται μία αποτελεσματικό το έγγραφο. Έχουμε και τον Σύρα Ρέγο από την Γκουε, παρακαλώ. Σύρα Ρέγο, η κυρία Σύρα Ρέγο από την Γκουε. Ευχαριστώ πολύ για μας ένας από τους μεγάλους προβληματισμούς ε, είναι ότι μπορούν ε, τα στοιχεία αυτά ε, να τα μοιραστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες και επομένως μας προβληματίζουν ζητήματα τα οποία αφορούν πληροφορίες σχετικά με το σεξουαλικό, θρησκευτικό, εθνικό προσανατολισμό των χωρών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην βάλουμε σε κίνδυνο ακόμα μεγαλύτερο πρόσφυγες ας πούμε μετανάστες π.χ. από το Σουδάν που ήδη αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Ε, και οπωσδήποτε πρέπει να κινούμαστε βάσει των διεθνών κανόνων. Επίσης, ε, ε, η διαμήραση πληροφοριών με ιδιώτες όπως είναι τα αεροπορικά, οι αεροπορικές εταιρείες, αυτό δεν μπορεί να μας βρει σύμφωνος. Θεωρώ ότι το άρθρο 32 της Συμφωνίας της Γενέβης ιδιαιτέρως αντιτίθεται σε τέτοιου είδους αρχές. Αναφέρει δε ότι με παραποιημένα ή όχι έγγραφα ταξιδίου άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται προστασίας πρέπει να την βρουν την προστασία αυτή. Επίσης ε, θέλουμε να είναι ε, ανοιχνεύσιμα άμεσα τα άτομα τα οποία έχουν δικαίωμα στην ε, διεθνή προστασία. Νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν με τον τρόπο αυτό να περιορίσουμε και με τέτοια μέσα να περιορίσουμε την είσοδο ανθρώπων, ανθρώπων λέω, Κοιτάξτε, ε, δεν είναι μηχανήματα, λέει ο Πρόεδρο, αυτοί που μεταφράζουν όταν μιλάτε. Είναι άνθρωποι, επομένω, να προσέχετε λίγο όσον αφορά την ταχύτητά σας. Ναι, ζητώ συγγνώμη, λέει η κυρία Σύρα Ρέγο. Συνεχίζω λοιπόν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διασφαλίζεται ε, το δικαίωμα στη διεθνείς μετακινήσεις, το δικαίωμα προστασίας ε, των προσωπικών δεδομένων και ε, βεβαίως δεν συμφωνούμε με το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι δικές μας θέσεις από την εισηγήτρια όταν έκανε τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Λοιπόν, δεν θέλετε δεν θέλετε κυρία Ματσόνα να πάρετε το λόγο. Ναι, είχα πει στην αρχή ότι δεν θα αντιδράσω. Παρ' όλα αυτά να πω ότι ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που άκουσα. Ενδεχομένως θα υπάρξουν κάποιε επιπλέον φραστικές διατυπώσεις έτσι, διαφορετικές έτσι ώστε να ε, ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσει των συναδέλφων. Λοιπόν, για το χρονοδιάγραμμα, η προθεσμία για τις τροπολογίες θα είναι 12 Νοεμβρίου. Μάλλον για την ψήφιση τους. 2 Νοεμβρίου, αν άκουσαμε καλά τον πρόεδρο, θα είναι για την υποβολή. μάλλον στη δεύτερη ολομέλεια του Νοεμβρίου θα ψηφιστεί. Λοιπόν, τώρα... Σχετικά με τις αιτήσει ασύλου, που είναι το επόμενο θέμα, η κυρία Βυσνιεύσκα είναι εδώ η συγκεντρία μας από το ECR. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Σχετικά με τον κανονισμό Eurodac, επιτρέπεται να τον συμβουλεύονται οι αρχές επιβολής του νόμου σε περίπτωση ποινικών αδεκημάτων βίων περιστατικών τρομοκρατικών επιθέσεων και άλλων τέτοιων περιπτώσεων και είναι πολύ σημαντικό εργαλείο στις εισαγγελικέ και ανακριτικές έρευνες. Υποβάλλουν λοιπόν, θα μπορούσαν να υποβάλλουν οι αστυνομικέ αρχές έτοιμα να συγκριθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα με εκείνα που αποθηκεύονται στην Κεντρική Τράπεζα Δεδομένων του Ντάκ, προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω πληροφορίε για την πρόληψη ε, ή την έρευνα τέτοιων αδικημάτων σαν αυτά που σας ανέφερα. Μιλούμε λοιπόν για την αναδιατύπωση του κανονισμού αυτού, αντικείμενο της οποίας είναι να παράσχει τη δυνατότητα στην Ελβετία και το Λίχτενστάιν ή μάλλον τις αστυνομικές τους αρχές λέει η ομιλήτρια και όχι τις ίδιες τις χώρες να μπορούν να συγκρίνουν τα δεδομένα που αφορούν στις δικές τους ερευνητικές υποθέσεις με τα δεδομένα που θα βρίσκονται στην Τράπεζα Δεδομένων Eurodac όταν προσπαθούν να ταυτοποιήσουν πρόσωπα που σχετίζονται με συγκεκριμένες τέτοιες περιπτώσεις κρουσμάτων, επιθέσεων, ερευνών κτλ. Είναι σημαντικό να μπορεί να συγκρίνει κανείς τα δεδομένα ιδιαίτερα των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η δική μου σύσταση, πρόεδρε, είναι να υποστηριχθεί η πρόταση αυτή και η έκθεση αυτή. Now we've heard. Λοιπόν, ακούσαμε την συγκέντρια, την κυρία Βυσνιεύσκα. Δεν είναι μόνο το πρωτόκολλο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Λίχτενστάιν, αλλά και της Νορβηγίας και της Ισλανδίας οι περιπτώσεις. Πρόκειται λοιπόν για πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των χωρών. που μπορεί να είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει ο Πρόεδρος, αλλά είναι εντός της Ευρώπης. Η κυρία Μετσόλα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης εκ μέρους του ΕΛΚ σε αυτό το θέμα. Ε, συμμεριζόμαστε την εισηγητρία στο σχέδιο της έκθεσής της για τα δύο πρωτόκολλα που θα προέκτηναν τις ε, διατάξεις επιβολής του νόμου για τις ε, τέσσερις αυτές χώρες μέσω διεθνούς συμφωνίας η οποία είχε ήδη ολοκληρωθεί προκειμένου τα στοιχεία ασύλου να, του Eurodac να ολοκληρωθούν. Με αυτό πλέον θα επιτρέψουμε στις αστυνομικέ αρχές των τεσσάρων αυτών χωρών να προβαίνουν σε σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχουν συλλέξει οι ίδιες με εκείνα που έχουν συλλέξει οι υπόλοιπε χώρες του Eurodac. Οι χώρε αυτέ λοιπόν και άλλες συνδεδεμένε χώρε θα, θα είναι σε θέση να ζητούν τέτοια σύγκριση. Μάλλον και οι χώρε μέλη θα μπορούν ε, αντιστοίχω να ζητούν το ίδιο α, ε, για τα σύγκριση δακτυλικών αποτυπωμάτων που έχουν γίνει από πλευρά των τεσσάρων αυτών χωρών. Θα έχουμε τις ρήτρε διαφύλαξης για τα προσωπικά δεδομένα και ελπίζω να έχουμε υιοθέτηση με απλή απλουστευμένη διαδικασία και ελπίζω επίσης να έχουμε θετική έκβαση και για τις δύο αυτές διεθνείς συμφωνίες. Η, κυρία Σάντος που επίσης είναι σκιώδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια για την παρουσίαση της ε, έκθεσής της. Περιέγραψε το περιεχόμενο του κειμένου που έχει συντάξει με ακρίβεια θα έλεγα. Πράγματι, οι τέσσερις αυτές χώρες θα αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία της ε, βάσης δεδομένων Eurodac για την ε, σύγκριση δακτυλικών αποτυπωμάτων σε περιπτώσεις ε, σοβαρών εγκλημάτων, τρομοκρατίας και βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να δώσει τη συγκατάθεσή του σε αντίστοιχα πρωτόκολλα. Ε, κάτι αντίστοιχο είχε γίνει παλαιότερα και με την ε, Δανία. Ε, πρόκειται για περιπτώσεις όπου η πρόσβαση αυτή δεν εξασφαλιζόταν μέχρι σήμερα, γι' αυτό και χρειάζεται να τροποποιηθεί ε, το ε, πρωτόκολλο. Δεν είναι κάποιο ακαθόδε θέμα, δεν είναι κάποιο θέμα στο οποίο μπορούμε να διαφωνήσουμε. Υπάρχει ευρύτατη συνένεση, γι' αυτό και εγώ νομίζω ότι δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε όσα είπε η συγγήτρια πάρα πολύ ωραία μας τα παρουσίασε. Εκτός μικροφώνου ο πρόεδρος. Represented here, so it'll be Mrs. Brickmont for the Greens. Η κυρία Βρυγκόν εκ μέρους των Πρασίνων. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Όλα υπόθηκαν όσον αφορά τα δύο θέματα που μας αφορούν εδώ στη μερίσια διάταξη. Ωστόσο, μια και είμαστε ε, ε, ανανεωμένοι κατά δύο τρίτα ε, εδώ, παρότι δεν είναι πολυπληθές το ακροατήριο, θέλω να πω ο, δύο λόγια σχετικά με την Eurodac, έστω και αν δεν μιλάμε για μια μεταρρύθμιση στο σύνολό της, παραμένουν κάποια προβληματικά ζητήματα που πρέπει να υπενθυμίσουμε, κυρίως το γεγονός ότι εμείς ως πράσινοι ε, υπενθυμίζουμε στο Συμβούλιο ότι θέλουμε να ε, ξεμπλοκάρει η συζήτηση για το ε, Δουβλίνο και ότι η μεταρρύθμιση της Eurodac θα πρέπει να εγγραφεί σε αυτή την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση την οποία θέλουμε εν είδη δέσμης να αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά τη Eurodac αυτό που μας προβληματίζει είναι η διεύρυνση της τακτικής στους παράτυπους μετανάστες που έχουν μπει νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εκεί θέλουμε να δούμε το θέμα της ε, χρησιμότητας μιας τέτοιας ε, διεύρυνσης. Επίσης, τη ε, μείωση της ηλικία από τα 14 στα 6 έτη για την λήψη αποτυπωμάτων. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται, θα εφαρμόζονται αρχές οι οποίες τρομάζουν τους ανηλίκους, ενώ θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της εξαφάνισης αυτών των ανηλίκων Τρίτον, ε, το θέμα του εγκλισμού ε, ε, και το σύστημα εγκλισμού δηλαδή έτσι ώστε να ληφθούν τα αποτυπώματα. Αυτό αποτελεί κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι υπερβολική, κυρίως ψυχολογική, υπερβολική δύναμη και βία ε, για την λήψη ε, των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη ευρύτερη μεταρρύθμιση. Από την ΚΟΕ δεν βλέπω. Έχει εγγραφεί μια συνάδελφος, αλλά δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος ε, σκιώδης. παρακαλώ λοιπόν την εισηγήτρια κυρία Βυσνιάσκη και αν θέλει να πάρει το λόγο. Δεν ξέρω αν θέλετε. Βέβαια μπορεί και αν θέλετε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, νομίζω ότι υπόθηκαν όλα όσα έπρεπε να υποθούν. Μιλάμε για την Ελβετία, την Ισλανδία, την Νορβηγία και το Λίχτενστάιν. Θέλω λοιπόν να δράξω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις, όλους τους συνεισηγητές και ελπίζω να μην υπάρξουν περαιτέρω τροπολογίες για αυτά τα δύο πρωτόκολλα γιατί ξέρετε ότι είναι μια τυπική διαδικασία οπότε μπορούμε απλώς να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας και να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Πολύ ωραία τα είπατε λέει ο Πρόεδρος. Ε, πράγματι η διαδικασία Συμβουλίου έχει ε, πολύ συγκεκριμένους περιορισμούς όσον αφορά τις ε, αρμοδιότητες τροποποίησης ε, από πλευράς του Κοινοβουλίου. Επομένως μετά την ε, επικοδομητική στάση που ακούσατε από όλες τις πλευρές να σας πω ότι οι τροπολογίες μπορούν να, να κατατεθούν έως 22 Νοεμβρίου, η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει 9 Δεκεμβρίου και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει τον Ιανουάριο του 2020. Νορβηγία, Ισλανδία. Για την Ελβετία και το ε, Λιχτενστάιν υπάρχει άλλη προθεσμία. Αυτά που σας είπα ε, ισχύουν για τις πρώτες δύο χώρες. 25 Οκτωβρίου, τροπολογίες, ψηφοφορία στην Επιτροπή 12 ή 11 Νοεμβρίου και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει στη δεύτερη Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Αυτά για απόψε. Σας ευχαριστώ όλους. Καλό σας βράδυ. Γεια.